Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Welcome back. Σωρίσατε και πάλι. Εντάξει με τα μικρόφωνα. Με ακούτε. Χθες ήταν μεγάλη μέρα Σήμερα θα είναι μια εξίσου μεγάλη μέρα, διότι πρέπει να προωθήσουμε ορισμένα θέματα, ξεκινώντας με το υπαριθμόν 8. Προτού όμως προχωρήσουμε στο 8, θα ήθελα να σας κάνω ορισμένε ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, σήμερα προ, την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας θυμίζω λοιπόν ότι πρέπει όσοι δεν έχουν την ηλεκτρονική κάρτα να την αναζητήσουν. Σε μία ώρα περίπου θα αρχίσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και το δεύτερο, όπως είπα χθε, το 14, το σημείο 14 έχει αναβληθεί, το οποίο σημαίνει ότι το 15 που αφορά την ακρόαση που θα έχουμε με ε, την Επιτρομάλστρομ για το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων που έγινε που θα γίνει στις 17 προβλέπεται στις 16 στις 16 στις 4 δηλαδή θα έχουμε ε, τον Επίτροπο Μάλστρομ γι' αυτό τώρα ερχόμαστε στο σημείο 8 που αφορά την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου της Σέγγεν στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Εδώ θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Κοέλιο υπό το φως των αποτελεσμάτων, των αξιολογήσεων και των επισκέψεων που έγιναν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η έκθεση συντάχθηκε με αντικείμενο να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να υιοθετήσει τη γνωμοδότηση ε, στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Θα μας μιλήσει ο κύριος Κοέλιο, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να έχετε υπόψη ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 14 Απριλίου. 14 Απριλίου για να εγκριθεί η έκθεση στη συνεδρίασή μας στη δεύτερη, τη 2 Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα λαμβάνει υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς, δηλαδή ε, τις διακοπές του Πάσχα, ε, το χρόνο που χρειάζεται για τη μετάφραση και θέλουμε ε, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια να γίνει πριν από το Συμβούλιο Τζάι. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να υποβάλουμε τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι εάν το Κοινοβούλιο έλαβε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες. Δεύτερον, κατά πόσο η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι έτοιμες να μπουν στο χώρο Σέγγεν. Η τρίτη είναι να συγκρίνουμε αυτή τη διεύρυνση Σέγγεν με την ε, τελευταία διεύρυνση Σέγγεν και τις διαφορές που υπάρχουν και επίσης να δούμε ποια άλλα θέματα σχετίζονται άμεσα με το θέμα μας. Πρώτον, λάβαμε τα έγγραφα. Ναι, πράγματι, το Συμβούλιο δεν συμπεριφέρθηκε καλά εξ αρχής. Προσπάθησε να αποφύγει τη συμμετοχή των βουλευτών στην διαδικασία αξιολόγησης. Εμείς αντιδράσαμε καλά οι δύο ενδιαφερόμενες χώρες, η Ρουμανία και Βουλγαρία, βοήθησαν με την ε, διαδικασία άρσης του απόρριτου χαρακτήρα των ε, εγγράφων. έτσι λάβαμε τις ε, κατάλληλες προφυλάξεις έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διαρροή πληροφοριών που να για την οποία αναφέρουμε εμείς ευθύνη. Εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα τη τελευταία έκθεση αξιολόγησης, εκείνη που σχετίζεται με την αξιολόγηση των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Λάβαμε άτυπα ορισμένα στοιχεία. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ως εισηγητή σας, και οι σκιώδεις και οι άλλοι μάλλον συντάκτες είδαμε in loco πώς έχουν οι προετοιμασίες. Μεταβήκαμε εκεί και είδαμε και τους ελέγχους στα σύνορα, πώς διενεργούνται δηλαδή. Άρα σε σχέση με τις πληροφορίες μπορώ να πω ότι λάβαμε τις πληροφορίες, θα λάβουμε και την τελευταία έκθεση το Κοινοβούλιο έχει όλες τις πληροφορίες για να τεκμηριώσει την άποψή του. Τώρα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες. Η απάντησή μου είναι ναι. Αυτό φαίνεται από όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης και από την επίσκεψή μας. Και όπως υπογράμμισα σε ορισμένες τομείς, αυτές οι χώρες είναι ακόμα πιο προετοιμασμένες από τις χώρες που είναι μέλη ήδη του χώρου Σέγγεν. Αυτό απορρέει από τις συνθήκες, δηλαδή ότι έχουν καλύτερο εξοπλισμό, πιο αποτελεσματικό αυτές οι χώρες και βεβαίως έγινε και μία πολιτική επένδυση από αυτές τις δύο χώρες έτσι ώστε να καταδείξουν ότι πληρούν όλους τους όρους προσχώρησης. Πώς συγκρίνω αυτή τη διεύρυνση με την τελευταία του 2007 όπου εννέα χώρες μπήκαν στο χώρο Σέγκε. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις. Δηλαδή το 2007 υπήρχε η πολιτική θέληση επαρκώς αιτιολογημένη να διευρύνουμε την ε, προσχώρηση μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2007 στην περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά σε ορισμένες χώρες υπήρχαν ορισμένα προβλήματα προς επίλυση, δηλαδή υπήρξαν πολλές ελλείψεις το 2007, κάτι το οποίο δεν επαληθεύεται σήμερα. Δηλαδή, σε σχέση με την εφαρμογή των κριτηρίων του Σέγγεν, όλα έχουν επιληθεί. Υπάρχουν μόνο μικρές λεπτομέρειες που θα πρέπει να επιληθούν, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το τι συνέβη το 2007. Τελευταίο ζήτημα, Πρόεδρε. Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται ακόμα με αυτό το ζήτημα. Δύο είναι τα ζητήματα. Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης σε σχέση με τα σύνορα Βουλγαρίας και Τουρκίας καταδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου προβλήματος. Υπάρχει μεγάλη μεταναστευτική ε, ροή, έκτακτη μεταναστευτική ροή μετά από την κατάσταση, την έκρηθμη κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και ζητήθηκε από τη Βουλγαρία να ορίσει ένα έκτακτο σχέδιο για να ανταποκριθεί στην έκτακτη μεταναστευτική αυτή ροή από την Τουρκία. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα. Εάν υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν βάσιμους φόβους σε σχέση με ανταπόκριση σε κατάσταση κρίσης, θα πρέπει να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις με έκτακτα σχέδια να υπάρχει ένας σύνδεσμος δηλαδή μεταξύ αυτών των σχεδίων και των επαληθεύσεων των κριτηρίων του Σέγγεν. Η Βουλγαρία δέχτηκε την αναγκαιότητα εκπλήρωσης αυτών των σχεδίων. Πολλά από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί, τώρα παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες και είμαι σίγουρος ότι η Βουλγαρία θα δώσει στους εταίρους όλες τις πληροφορίες που τις ζητήθηκαν. Ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με αυτό είναι η αποτίμηση του Σέγγεν, δηλαδή η αποτίμηση των εκθέσεων. Υπάρχουν θέματα που δεν πρέπει να διασυνδέονται μεταξύ τους. Εμείς έχουμε αρχίσει τη συζήτηση για το σύστημα αξιολόγησης του χώρου Σέγγεν και αυτό που είχα πει σε σχέση με το θέμα Σέγγεν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Δηλαδή άλλοι κανόνες για τις υποψήφιες χώρες και άλλοι κανόνες να ισχύουν για τα μέλη του Σέγγεν. Όταν αξιολογούμε για το κατά πόσο οι χώρες συμβαδίζουν ή όχι με τα κριτήρια του Σέγγεν, όλοι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το ίδιο κριτήριο. Δηλαδή είτε κάποιος, κάποια χώρα είναι υποψήφια είτε βρίσκεται στο χώρο Σέγγεν. Και επ' αυτού θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρωτοβουλία ορισμένων κρατών μελών στο Συμβούλιο που θέτουν ένα αμφιβόλο τη νομική βάση που και που θέλουν να αποσυρθεί το Κοινοβούλιο από τη συναπόφαση του νέου συστήματος ε, Σέγγεν. Αυτό σημαίνει ότι υποβαθμίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να επιδράσουμε επί αυτής της νομοθεσίας. Όπως σας είχα πει, με βάση το πρώτο σύστημα αποτίμησης τότε δεν προβλεπόταν η συναπόφαση και εμείς απορρίψαμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ζητήσαμε από την Κομισιό να υποβάλει ένα νέο σχέδιο. Τώρα που η Επιτροπή το δέχτηκε και εφόσον νομική βάση προϋποθέτει τη συναπόφαση υπάρχουν κράτη που θέλουν να προκαλέσουν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου σε σχέση με την θέση ορισμένων κράτων μελών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία που προσπαθεί να κρατήσουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως είχε προταθεί αρχικά σε σχέση με θέματα συναπόφασης. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο για την έκθεσή σας. Και πριν δώσω το λόγο τη Επιτροπή, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Προεδρία. Η Προεδρία του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, πείτε μας το όνομά σας. Καλημέρα. Τι Μέιλ είναι το όνομά μου. Και προεδρεύω την ομάδα του Συμβουλίου που αξιολογεί τη Συμφωνία Σέγγεν υπό την αιγίδα της Προεδρίας και είμαστε και υπεύθυνοι για το θέμα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, ότι η Προεδρία θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα ε, το θέμα του Σέγγεν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις θέλουμε να μπουν η Ρουμανία και η Βουλγαρία το συντομότερο δυνατόν στο χώρο Σέγγεν. Όπως γνωρίζετε, το Δεκέμβριο του 2010 καταρτίστηκε η έκθεση χώρας για τη Ρουμανία και εγκρίθηκε η έκθεση αυτή. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, δεν έγινε το ίδιο, το Δεκέμβριο δηλαδή, αλλά θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία το Μάρτιο, μπορέσαμε συγγνώμη, να επαναλάβουμε τη διαδικασία το Μάρτιο και αξιολογήσαμε την κατάσταση για τη Βουλγαρία και πάλι το Μάρτιο με θετικά συμπεράσματα. Το σχέδιο έκθεσης το υποβάλαμε τον Απρίλιο, ούτως ώστε αρχές Μαΐου ελπίζουμε να εγκριθεί. Έχω ξαναπεί ότι η Προεδρία γνωρίζει ότι το θέμα αυτό έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχουν εγγυήσει για την ασφάλεια του χώρου Σέγγεν και οι χώρες που μπαίνουν στον χώρο Σέγγεν θα πρέπει να διασφαλίζουν αυτά τα θέματα. Η συμφωνία στο Συμβούλιο πρέπει να είναι με ομοφωνία. Το Φεβρουάριο στο Συμβούλιο ΔΕΗ συζητήσαμε το θέμα αυτό και φάνηκε ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν ήταν σίγουρα ότι μπορούν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως η Προεδρία θα προσπαθούσε να οδηγήσει σε κάποια βεβαιότητα όλα τα κράτη-μέλη σχετικά με τις δύο αυτές χώρες. Οι προσπάθειες και των δύο χωρών, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, ε, είναι αξιέπαινες γιατί έχουν καταβάλει και οικονομικές προσπάθειες και άλλες προσπάθειες και οι δύο χώρες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια λύση για να επιβραβευθούν τουλάχιστον για τις προσπάθειές τους. Και ο στόχος είναι το να γίνουν πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Τώρα η κυρία Τζοάννα Τέμπλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν θέλει η Επιτροπή το λόγο, ξεκινάει η συζήτηση. Τα μέλη της Επιτροπής μας. Σημειώνω Ποιο ζητάει το λόγο. Yes. We're getting started. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κυρία Γιωτόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο, για τη δουλειά που έκανε και για το σχέδιο έκθεσής του. Και θα ήθελα να πω ότι στηρίζω την θέση του και τα συμπεράσματά του και παρότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στις δύο τελευταίες εκδοχές του κειμένου. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Κοέλιο διότι διατυπώσατε την άποψη ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Βουλγαρία σε θέματα ασφάλειας από ότι ορισμένα παλαιότερα κράτη-μέλη κατά την ένταξή τους. Θα ήθελα να τονίσω την διαφωνία μου για την ανάμειξη κριτηρίων αξιολόγησης, το μηχανισμό αξιολόγησης του κεκτημένου Σέγγεν και την αξιολόγηση των μηχανισμών συνεργασίας και επαλήθευσης. Υποστηρίζω τη δημιουργία νέου συστήματος εξέλιξης Σέγγεν με σαφέστερους κανόνες και συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν όλα τα κράτη-μέλη. Όμως η δημιουργία του νέου μηχανισμού θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από την τύχη που επιφυλάσσουμε στη Βουλγαρία και Ρουμανία και δεν θα πρέπει να φύγεται η ένταξή τους στο χώρο Σέγγεν. Πρέπει να αποφύγουμε το να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα νέα κρατημέλη και τα παλαιά κρατημέλη. Επίσης θέλω να τονίσω ότι το προβλήμα που βλέπουμε τώρα μεταξύ Ιταλίας και άλλων κρατών μελών δείχνουν τη σημασία που έχουν όλα αυτά τα θέματα για το χώρο Σέγγεν και ελπίζω ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τις δύο χώρες και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Βλέπουμε μια θετική έκθεση και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη Βουλγαρία και Ρουμανία στο χώρο Σέγγεν. Ελπίζω ότι οι υπολοιπόμενες διαδικασίες στο Συμβούλιο θα γίνουν με βάση ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, ούτω ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης, Νομίζω ότι έχει κέρια σημασία οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο χώρο Σέγγεν να συνεχίσουν να τηρούνται και μετά την ένταξη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες σήμερα συμπεριλαμβανομένων των χωρών που αντιμετωπίζουν την πίεση από τη μετανάστευση. Η διαδικασία Σέγγεν συνεχίζει να τονίζει την ιδέα ότι ε, παραμένει μεν κάθε κράτος μέλος υπεύθυνο για τα εξωτερικά του σύνορα, αλλά ταυτόχρονα είναι όλο και περισσότερο σαφές ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν κοινό μέλημα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο από το πνεύμα ε, του Σέγγεν. Δυστυχώς δεν είναι απόλυτα σαφές για όλους μας, για όλες τις χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω συμμετάσχει στην αξιολόγηση των εκθέσεων και γι' αυτό είναι δύσκολο να σχολιάσω λεπτομερώς τα θέματα, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να κάνω γενικές παρατηρήσεις για αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο, ο οποίος όπως πάντοτε έκανε ένα θαυμάσιο έργο και θα ήθελα κυρίως να σας ευχαριστήσω επειδή αγωνιστήκατε για να υπάρχει πρόσβαση ε, των Ευρωβουλευτών όσον αφορά τις εκθέσεις αυτές. Μέχρι τώρα ήταν γελίο το γεγονός ότι δεν είχαμε πλήρη ε, πρόσβαση ε, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πάνω στα θέματα. Για μένα όμως το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουμε πλέον διπλά μέτρα και σταθμά και δεν πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προτού προσχωρήσουν στο Σέγγεν από ό,τι κάναμε με τα άλλα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν δίκαιο, θα ήταν άδικο. Γι' αυτό με τα σας διαπιστώνω ότι ο εισηγητής καταλήγει ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια για πλήρη προσχώρηση ε, στο Σέγγεν ούτε για τη Ρουμανία ούτε για τη Βουλγαρία διότι έχουν συμμορφωθεί πλήρως και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει πολύ ευαίσθητα σύνορα κυρίως μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας θα μπορούσαμε να προβλέψουμε να υπάρχει ε, αυξανόμενη παράνομη μετανάστευση και οι συνοριακοί φύλακες θα πρέπει να λειτουργήσουν πολύ καλά σε αυτά τα σύνορα. Σημαντικό είναι λοιπόν να εκπαιδεύονται σωστά, να γνωρίζουν πώς να υποδέχονται τα άτομα τα οποία χρειάζονται διεθνή προστασία. Και επίσης ε, μπορούμε να προβλέψουμε την ε, αυξανόμενη ανάγκη διερμηνέων που θα πρέπει να είναι παρόντες στα σύνορα. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να σκεφτούμε να συμμετάσχει και η Frontex, η Frontex στην εκπαίδευση των συνοριακών φυλάκων και των διερμηνέων κυρίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι ουσιαστικό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ώστε τα προγράμματά μας ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ μας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν μέχρι τώρα και ευχαριστώ και πάλι κύριε Κοέλο. Κύριε Σέντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα όπως και οι άλλοι προλαλήσαντες να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για το έργο που επιτέλεσε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα όμως να τον ευχαριστήσω και για την άλλη έκθεση που αφορά την εφαρμογή ε, του κεκτημένου του Σέγγεν. Θα ήθελα επίσης να κάνω ορισμένες άλλες παρατηρήσεις, τις οποίες όμως ανέφερε ο κ. Κοέλιο. αυτή είναι ίσως η αιχμή του δόρατος αυτού του αγώνα που γίνεται και που γίνεται μια προσπάθεια να αφαιρεθεί μέρος των ευθυνών μας από αυτή τη διαδικασία αποφάσεων. Τα άλλα θεσμικά όργανα μέχρι τώρα προσπάθησαν να μας βάλουν σε μια ε, κατάσταση εμπλοκής ε, πάντοτε αναφερθήκανε ε, ισχυρισμοί, επιχειρήματα για να καθυστερήσει αυτή η έκθεση. Ο εισηγητής μας όμως κατέδειξε ότι μπόρεσε να αγωνιστεί, ότι μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή την έκθεση και ήταν ικανός να ζητήσει την κατάλληλη στιγμή να γίνουν επισκέψεις στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να δούμε επιτόπου ποια ήταν η πραγματική κατάσταση. Κανείς τώρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει όλα αυτά που έγιναν ορισμένα πράγματα υπήρξαν απόλυτα σαφή. Μερικές φορές έχουμε ικανότητες μεγαλύτερες από άλλες χώρες που ήδη ανήκουν στο Σέγγεν. Γι' αυτό θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τον εισηγητή μας και για αυτή την έκθεση αλλά και για τις επόμενες εκθέσεις που θα αφορούν πάντοτε ε, το Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ με τη σειρά μου τον εισηγητή κύριο Κοέλο για τη θαυμάσια εργασία που έκανε, μια θαυμάσια εργασία ουσία που βασίστηκε στην προετοιμασία των δύο χωρών. Ακούσαμε η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμε να εισχωρήσουν το Σέγγεν. Οι εκθέσει τη Επιτροπή ΕΒΑΛ έδειξαν ότι δεν υπάρχει λόγο να σταματήσει η εισδοχή αυτών των χωρών. Άλλωστε είδαμε ότι δύο χώρε έλαβαν μέτρα που ξεπερνούν εκείνα τα οποία είχαν λάβει τα ε, κράτη που ήδη ανήκουν στον χώρο Σέγγεν. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσω για τα εξή. Αυτό το οποίο προτείνει ο εισηγητή, τα ειδικά σχέδια είναι θετικά, διότι σύμφωνα με τα πορίσματα του ΣΕΒΑΛ και του εισηγητή, εμεί δεν εμποδίζουμε την προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν, αλλά μάλλον επιτρέπουμε την είσοδό του με τη δυνατότητα να παρακολουθούνται ειδικά μέτρα. Δεύτερον, είναι κατανοητό το γεγονό ότι η Επιτροπή Αξιολόγηση να έχει ορισμένε επιφυλάξει όσον αφορά την μεταναστευτική πίεση. Αυτή είναι μια συνεχή πρόκληση που αντιμετωπίσουν όλε οι νότιε χώρε στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρώπη. Οι βουλγαρικέ αρχέ το γνωρίζουν και ελπίζουμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί. Οποιοδήποτε αίτημα που αφορά αυτό το θέμα θα πρέπει όμω να τοποθετηθεί σε όρια και να μην είναι πρόσχημα για να καθυστερήσει η προσχώρηση της Βουλγαρίας στο, στο χώρο Σέγγεν. Τρίτο, Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι τα συμπεράσματα να είναι τα δικαιότερα. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο στη χώρα μου. Η προσχώρηση στο Σέγγεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο μιλάει, αν θέλετε. Είναι και το σύμβολο τη Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε στου πολίτε μα ναι, ε, ναι, μεν πληρείτε τα κριτήρια, αλλά για πολιτικού λόγου δεν μπορείτε να ε, προσχωρήσετε στο Σέγγεν. Αν το κάνουμε αυτό, τότε αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά και Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Τέλο, είναι σημαντικό να δούμε και πάλι το σύστημα αξιολόγηση του Σέγγεν, διότι μερικέ φορέ είμαστε πολύ αυστηροί με του νέου, αλλά όχι με του παλιού που έχουν εισχωρήσει. Στο μέλλον πρέπει οπωσδήποτε οι εκθέσει αξιολόγηση των διαφόρων κρατών μελών να βασίζονται στα πραγματικά γεγονότα. Δεν μπορούμε να έχουμε εκθέσει οι οποίε είναι δύσκολε και να τις βάζουμε στα σιρτάρια και να τα κλειδώνουμε. Η έκθεση που θα παρουσιάσει ο κ. Σκοέλο ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση και εκ των τον ευχαριστώ και σύμφωνα με αυτά πιστεύω για μία ακόμη φορά ότι θα προσφέρουμε μεγάλη υπηρεσία και στην Ευρώπη και στους πολίτες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους όσους ευχαρίστησαν τον κύριο Κοέλο, συντάκτη της έκθεσης. Κατά τη γνώμη μου, κατόρθωσε να, να συνδυάσει δύο σημαντικές λεπτομέρειες στην προσέγγιση του σε αυτό το πολύ περίπλοκο θέμα που έχει σχέση με την εισδοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο Σέγγεν. Υπήρξε και πολύ επαγγελματίας και πάρα πολύ τίμιος. Υπενθύμησε σε όλους μας ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το ίδιο στυλ, αν θέλετε. Μιλώντας λοιπόν για αυτές τις δύο χώρες, καταλήγουμε ομόφωνα στο εξή συμπέρασμα. Αυτές οι χώρες είναι έτοιμες. Σε άλλες ε, εκδοχές είχε υποστηριχθεί με άλλα κριτήρια, με άλλες εντυπώσεις ε, που υπήρχαν όταν έγιναν οι επισκέψεις ε, στα σύνορα των δύο χωρών. Αλλά η πραγματικότητα μας ζητεί όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, στους Ευρωβουλευτές και στους εισηγητές, αλλά και στα άλλα θεσμικά όργανα, να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτό το όραμα για την αναπόφευκτη προσχώρηση των δύο αυτών χωρών στο Σέγγεν. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος από ηθική άποψη για τις κοινωνίες, για τους πολίτες αυτών των χωρών. Κανείς δεν είναι σε θέση ούτε τα ΜΜΕ ούτε η πολιτική να αποτρέψουν κάποιο σκεπτικισμό στην Ρουμανία και τη Βουλγαρία εάν μετά τον Ιούλιο ή μετά τον Σεπτέμβριο υπάρχει ακόμη αναβολή. Βεβαίως δεν χρειάζονται αυτές οι χώρες ούτε χριστουγεννιάτικο δώρο ούτε καλοκαιρινό δώρο. Χρειάζονται αξίωση των προσπαθειών τους. Στη χώρα μου, στη Βουλγαρία, πάνω από 130 ε, εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν σε εξοπλισμό, σε πλοία, σε ελικόπτερα, σε εξοπλισμό παρακολούθησης, σε μηχανισμούς, προετοιμασίες διαφόρων ειδών. Η ικανότητα των αρχών, των συνοριακών φυλάκων, των αξιωματούχων στα σύνορα και στην συνοριακή ζώνη, ήδη αυτή η ικανότητα είναι πολύ υψηλή και αυτό το είδαν όσοι επισκέφθηκαν τέλη Μαρτίου τη χώρα. Τι άλλο πρέπει να αναφέρουμε σήμερα. Υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον στο κείμενο του κυρίου Κοέλο, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση ε, μεγάλη μεταναστευτική πίεση μετά την πρίλη προσχώρηση, η Επιτροπή Εξολόγηση καλεί την Βουλγαρία να ετοιμάσει ένα πακέτο συνοδευτικών μέτρων. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Ούτε να εκλειφθεί ως προσπάθεια να προσθέσουμε κάτι το καινούριο στα ήδη γνωστά κριτήρια που υπάρχουν για την εκτίμηση της συμπεριφοράς μιας χώρας η οποία θα προσχωρήσει στο Σέγγεν. Αλλά πρέπει να κλειφθεί ως μια ευελιξία που σε περίπτωση δυσμενών γεγονότων θα ενεργοποιηθεί. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της, του Συμβουλίου, μιλάμε για την ευαισθησία μεταξύ, ε, των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας ε, σας βεβαιώνω ότι αυτή η ευαισθησία βασίζεται σε ιστορικές και συναισθηματικές ρίζες. Συνεπώς πρέπει ορισμένα πράγματα να τα κατονομάζουμε σωστά, να τους δίνουμε το σωστό του όνομα σήμερα. Παράλληλα με αυτές τις προσπάθειες για να προσχωρήσουν αυτές οι δύο χώρες στο Σέγγεν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε ίσως να εστιάσει πάνω στα ε, προβλήματα που δεν έχουν λυθεί μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνία επανεισδοχής, δηλαδή τι συμβαίνει μεταξύ Τουρκίας και των γειτόνων της. Διότι επειδή η συγκέντρωση πιθανών μεταναστών από τους γείτονες, ε, ακόμα και από το Ιράκ, θα, θα αποτελέσει μέρος της εικόνας, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνε η Βουλγαρία και η Ρουμανία για αυτά τα πιθανά γεγονότα. Λέγοντας λοιπόν ότι ορισμένα προβλήματα απομένουν ε, και θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Σήμερα ε, συμφωνούμε με εκείνους που μας είπαν τα καλά μαντάτα ότι δύο χώρες είναι έτοιμες για να προσχωρήσουν ε, στο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Ευχαριστώ, κυρία Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και διότι ε, ε, με αξιοπρέπεια σώζει τη φήμη του Κοινοβουλίου ε, Έχουμε δει ότι υπήρχαν πολλά εμπόδια όσον αφορά ε, ε, τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφόρηση και σε έγγραφα σχετικά με τις αξιολογήσεις και νομίζω ότι για όλους μας ε, ήταν ένα θέμα που μας έφερε σε δύσκολη θέση έναντι Βουλγαρίας και Ρουμανίας και νομίζω ότι πραγματικά τίθεται θέμα αξιοπρέπειας για την αντιμετώπιση μας. Τώρα οι πολίτες της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανία νιώθουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε προς την κατεύθυνσή του. Με το άνοιγμα των συνόρων ε, νιώθουν κάτι περισσότερο. Και με το άνοιγμα των συνόρων για την Πολωνία και την Τσεχία το 2007 πάλι κατάλαβα ότι οι πολίτες ένιωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζουν ε, τις χώρες αυτές. Θυμάμαι ότι ήμουν στην ε, Τσεχία όταν άνοιγαν τα σύνορα για την Τσεχία και θυμάμαι ότι άκουσα στο ραδιόφωνο ε, σχετικά με τα μέτρα τα οποία ο τοπικός υπουργός ε, στην ε, συνοριακή περιοχή ε, στα σύνορα με τη Γερμανία ανακοίνωνε μέτρα για να μην έρθουν οι κλέφτες και διαδίκτες ε, από την Τσεχία. Έλεγε φτιάξτε καλύτερους φράχτες, κλειδώνετε τα σπίτια σας. Υπήρχε μια πραγματική ιστερία εκείνη την εποχή και γι' αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε τα, τα θετικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Παρότι η δική μου ομάδα για τα θέματα της μετανάστευση έχει διαφορετική εικόνα από ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου για τα θέματα της ε, μετανάστευση. Και για τη Βουλγαρία θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψη σα γενικά για το πακέτο αυτό. Και κάτι που επίσης θεωρώ σημαντικό θα ήθελα να το τονίσω προς τον κύριο Κοέλιο, είναι να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και το λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί υπάρχει αυτή η τάση να κατευθυνθούμε προς μια Ευρώπη που θα αποτελεί τον πυρήνα και γύρω-γύρω τα υπόλοιπα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να το επιτρέψουμε αυτό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Χρειαζόμαστε τους ίδιους κανόνες, τους ίδιους περιορισμούς και να εφαρμόζονται το ίδιο οι κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη. Να μην έχουμε ένα πυρήνα και άλλες χώρες στο περιθώριο. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι ε, ε, έχουμε τη δυνατότητα και την υποχρέωση να λάβουμε ενεργά μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα το έχουμε αποδείξει και χάρη στον συνάδελφο Κοέλιο έχουμε κάνει και πολύ σωστό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να επαναλάβω τη δήλωση που έκανε η ομάδα μας στην πρώτη συζήτηση για το θέμα ότι υποστηρίζουμε πλήρως όλες τις προσπάθειες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να μπουν στον χώρο Σέγγεν. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κοέλιο για το έργο του. Όχι μόνο πριν από την πρώτη συζήτηση, αλλά και τώρα, κατά την ε, τελευταία αυτή περίοδο, με την οργάνωση της ε, επίσκεψης στις χώρες αυτές. Η ομάδα μας ε, δεν συμμετέσχει αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα συμπεράσματα. Επίσης υποστηρίζουμε την τροπολογία που υπέβαλε ο κύριος Κοέλιο στην αιτιολογική σκέψη 4 και ε, χαιρετίζουμε τη νέα έκθεση. Η τροπολογία αυτή είναι πολύ σημαντική. Εποφελούμενη της παρουσίας της Προεδρίας του Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μας ε, σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. όταν τελικά μου δόθηκε πρόσβαση στην έκθεση αξιολόγησης, δοκίμασα μια διπλή ε, έκπληξη. Γιατί να υπάρχει μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία για να έχουμε πρόσβαση στην έκθεση αξιολόγησης. Διαβάζοντας την έκθεση, διαπιστώνω ότι δεν χρειαζόταν τόσο πολύπλοκη διαδικασία και ελπίζω ότι στις μελλοντικές προσπάθειες διεύρυνσης του χώρου Σέγγεν δεν θα επαναληφθεί αυτή η διαδικασία. Και ως ε, Ευρωβουλευτής από μια χώρα που μπήκε στο χώρο Σέγγεν το 2007 υποστηρίζω και τις συγκρίσεις που κάνει ο κύριος Κοέλιο με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εκείνη την εποχή και με τις διαδικασίες που ακολουθούνται τώρα για τη Βουλγαρία και Ρουμανία. Και πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλή θέση η Βουλγαρία και η Ρουμανία για να μπουν στον χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σκόβατσεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του, διότι η έκθεση αυτή ακριβώ υποδεικνύει αυτά που χρειαζόμαστε στο χώρο Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Πρέπει η διαδικασία για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να ολοκληρωθεί με την ίδια διαδικασία με την οποία ξεκίνησε. Ήδη από το 2007 είχαμε πει ότι αν οι δύο χώρε πληρούν τι προποθέσει, θα μπουν στο χώρο Σέγγεν στι αρχέ του 2011. Αυτό είναι ήδη γεγονό, διότι πληρούνται ήδη τα κριτήρια. Οτιδήποτε άλλο πέραν αυτών των αρχικά κατριτισμένων κριτήριων, είναι πολιτικού χαρακτήρα και ενδεχομένως εσωτερικού πολιτικού χαρακτήρα σε διάφορα κράτη-μέλη. Έναντι αυτών των βραχυπρόθεσμων ε, σκέψεων πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα την αντιμετώπιση ε, των κινδύνων στα εξωτερικά μας σύνορα, ιδιαίτερα τις απειλή από την ε, μετανάστευση. Αυτό είναι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η κρίση αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και στη Μάλτα. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για να συζητάμε νέου κανόνε, θα πρέπει να είναι κανόνε που θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, και τα παλαιά και τα νέα κράτη-μέλη. Το να είναι κανεί μέλο στο χώρο Σέγγεν δεν είναι κάτι το οποίο έχει στατικό χαρακτήρα. Πρέπει να είναι κάτι που αξιολογείται συνεχώ για να μπορούμε να αξιολογούμε τι νέε προκλήσει. Όταν οι χώρε μα είναι μέλη του χώρου Σέγγεν θα πρέπει να διατηρούν υψηλά πρότυπα και όχι να επαναπαύονται. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν κάνει το, την προσπάθεια που έπρεπε. Τώρα έχουν, έχουν καταρτήσει προγραμματισμό για ειδικέ ε, καταστάσει και μάλιστα και προγραμματισμό που δεν είναι τμήμα των κριτηρίων για την ένταξη στο χώρο Σέγγεν. Είναι κάτι το οποίο ε, απαιτείται από όλε τι χώρε ε, που βρίσκονται ε, στην πρώτη γραμμή, τι χώρε που πρέπει να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την έκθεση του εισηγητού και ε, μετά από τα συμπεράσματά τους από την επίσκεψη ε, στον εύξηνο πόντο ε, διαπιστώσαμε διαπίστωσαν και ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής και άλλοι τον τρόπο με τον οποίο διαφυλάσσουν τα εξωτερικά σύνορα τα θαλάσσια σύνορα προς τον εύξηνο πόντο η Βουλγαρία και η Ρουμανία και θα θέλαμε την ίδια φύλαξη να εξασφαλίζουμε και σε όλη τη φύλαξη των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου ομιλητέ να ζητούν το λόγο. Ήδη ακούσαμε αρκετέ παρεμβάσει. Ήταν μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα με πολλούς ομιλητές, όχι μόνο από τις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά και από συναδέλφους από όλες τις χώρες. Κύριε Κοέλη, νομίζω τώρα θα έχετε το χρόνο να σκεφτείτε όλα αυτά τα σημεία που αναφέρθηκαν. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω, απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τα, για τα καλά σχόλια του συναδέλφους και θα ήθελα να σας πω ο, το προθεσμίες που έχουμε ορίσει. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη γνωμοδότησή του πριν από τη συνάντηση του Συμβουλίου και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το Κοινοβούλιο είναι φωνή των πολιτών και θα πρέπει να γνωμοδοτήσει πριν από το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι κλείσαμε επί του παρόντος και πάλι σας θυμίζω ότι μέχρι τις 14 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα πρέπει να έχετε υποβάλει τις τροπολογίες σας, έτσι ώστε στις 2 Μαΐου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης. Τώρα νομίζω ότι έχουμε στις 10 μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ήθελα να πω ε, ότι θα πρέπει να διακόψουμε μάλλον για 10 λεπτά, γιατί πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να ψηφίσουν δεν παρευρίσκονται. Στις 10 ακριβώς θα αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Ε,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

Είμαστε έτοιμοι, έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Επαληθεύστε ότι έχετε την κάρτα σας. Για να προχωρήσουμε. Έχουμε το θέμα της ψηφοφορίας για τον ε, κατάλογο ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου. Η κυρία Τάνια Φαζόν είναι η συγγήτρια που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ο κύριος Ένσιου λοιπόν μπορεί να μας κάνει μια παρουσίαση ή αν δεν θεωρείται ότι είναι απαραίτητο μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Εγώ θα σας πω ποιες είναι οι τροπολογίες που έχουμε. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις. Τώρα τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 6. Ναι, είναι συμβιβαστική τροπολογία για το 6α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το τροποποιημένο κείμενο ψήφι υπέρ. Α, ναι, ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουμε, ναι, ναι, ναι. Ναι, θα ψηφίσουμε μία επιπλέον ψήφο για τους σοσιαλιστές, εντάξει. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας υπέρ μία ψήφος κατά. 29. 29 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Εγκρίνεται. Με βάση τις τροπολογίες, η κυρία Φαζόν θα αρχίσει συζητήσεις με το Συμβούλιο για να καταλήξουν σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση αν αυτό είναι δυνατόν. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι το σημείο 10 και έχουμε μία ώρα και 15 λεπτά για μία μίνι ακρόαση που αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια ακρόαση εμπειρογνωμόνων και την παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως της συναδέλφου Σόνια Αλφάνο. Ελάτε εδώ στο βήμα κυρία Αλφάνο για να παρουσιάσετε την έκθεση και έχουμε μία ώρα και ένα τέταρτο για να ακούσουμε και τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αποτελεί θέμα της ε, επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ε, να κάνουν μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό και αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ήταν ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν διάφορες ακροάσεις για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Αλφάνο, η συγγήτριά μας, θα μας παρουσιάσει και τους εμπειρογνώμονες που έχουμε για το θέμα αυτό. Κυρία Αλφάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν μπω στην ουσία του σχεδίου έκθεσης θα ήθελα να σας μιλήσω για τη μεθοδολογική μας πορεία. Πέραν από αυτή την πρόταση Υπάρχει και σωρία άλλων που δεν έχουν εισαχθεί στο κείμενο για λόγους χώρου, αλλά θα μπουν μέσω τροπολογιών. Είναι λοιπόν απότοκες μίας συνεργασίας με τους φορείς, υπηρεσίες, εμπειρογνώμονες, αστυνομικές δυνάμεις, με τα θύματα και το οικογενειακό περιβάλλον των θυμάτων, καθώς και με αρχές της δικαιοσύνης. Στις 29-30 Μαρτίου ορίστηκε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν 50 δικαστές που προέρχονταν από 18 διοικητικά τμήματα καταπολέμησης της μαφίας, αλλά είχαμε και έναν εισαγγελέα από την Ισπανία, έναν Καναδό δικαστικό και άλλους εισαγγελείς. Μπορώ να πω, χωρίς κανένα φόβο μήπως διαψευστώ, ότι... Κυρία Αλφάνο, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, θα ήθελα να επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα για να μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Αλφάνο. Σας παρακαλώ πολύ. Όποιος δεν θέλει ας αποχωρήσει. Έλεγα λοιπόν ότι μπορώ να πω ότι η Ιταλική πύρα αποτελεί ένα πρότυπο που θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι η, η Ιταλία είναι η χώρα η οποία κατά πολλά άρδινε τη μαφία, ξεκινώντας από δικαστές, δημοσιογράφους, οικογένειες θυμάτων και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ισαγγελέα μετά την ακρόαση της 29ης Μαρτίου, ο οποίος ε, μας εξήγησε και θα μας εξηγήσει ορισμένα τεχνικά μέτρα εγώ θα ήθελα να σας πω γιατί η έκθεση έχει ύψιστη σημασία και θα εξακολουθήσει να έχει και στο μέλλον. Θα ήθελα να να σταθώ στους λόγους για τους οποίους έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε για να προβάλλουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο από πολιτικής πλευράς. Θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Χαίρομαι που είμαι η συγγήτρια αυτής της έκθεσης και για προσωπικούς λόγους, αλλά γιατί η πολιτική μου εντολή σχετίζεται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα πλαίσια της καταπολέμησης της Ιταλικής μαφίας. Πρέπει να γνωστοποιήσω αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη σκέψη και η πιο σημαντική είναι ότι θα πρέπει να σταθούμε στις επιπτώσεις του οργανωμένου έγκληματος στη ζωή των πολιτών. Το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος διεισδύει στον κοινωνικό ιστό. Σκεφτείτε πόσα χρήματα δαπανώνται σε επίπεδο τοπικής ε, διοίκησης ή εθνικής για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα το οποίο μολύνει επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο και μολύνει το περιβάλλον καθώς και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ε, κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας. Δεν είναι ένα θέμα λοιπόν που οριοθετείται επακριβώς. Επειδή έχει διεισδύσει η μαφία στον ευρωπαϊκό ιστό, μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Πρόκειται για παράλογες διαστάσεις που διεισδύουν στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό και πλήττει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα με όλο ένα και μεγαλύτερη εθνική και ευρωπαϊκή σημασία αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Δυστυχώς υπάρχουν καλές προθέσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν με συγκεκριμένα αντίμετρα. πολλές φορές εξουσιοδοτούμε αυτό το έργο στην αστυνομία ή στους δικαστικούς που θα πρέπει να δώσουν δονκιχωτικές μάχες για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα. Η... Αυτό αφορά και τους πολίτες. Η θέση των πολιτών είναι η ίδια. Διότι όσοι έμποροι καταπολεμούν ή γνωστοποιούν αυτό το έγκλημα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουν περιορισμένη ισχύ. Όπως είπε ο Τζοβάνι Μαλφαλκόνε, ο οποίος σκοτώθηκε από την μαφία στις 23 Μαρτίου του 1992, δυστυχώς η οικονομική δραστηριότητα της μαφίας είναι ένα πάγιο φαινόμενο και θα πρέπει οι όλα τα θεσμικά όργανα να καταπολεμήσουν αυτό το ιδεχθές φαινόμενο. Πρέπει να τιμήσουμε τον δικαστή Μανφαλκόνε και το λεγόμενό του και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκριμα. Δεν έχει σύνορα, δεν έχει σημαία, δεν έχει πολιτικό κόμμα η μαφία. Και γι' αυτό όλοι οι βουλευτές θα δέχονταν τις προτάσεις του Τζοβάνι Φαλκόνε. Γι' αυτό θα πρέπει να αποστείλουμε συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία να μην την χάνουν πολλαπλών ερμηνεών. Δεν μπορούμε να νικήσουμε το οργανωμένο έγκλημα εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ερευνητικές και ανακριτικές αρχές που να μπορούν να λειτουργήσουν με τα επαρκή μέσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει συγκεκριμένη ευθύνη έναντι των πολιτών της, γι' αυτό θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να παράγουν απτά αποτελέσματα. Η Europol με τις αιτήσιε εκθέσεις της αναγνωρίζει εδώ και χρόνια την έκδηλη παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρω... στον ευρωπαϊκό ιστό. Άρα έχουμε στρέβλωση των αγορών και καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Παράλληλα, και πέρα από αυτή την ε, έκθεση της Europol και την περιγραφή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα χαλαρή. Το 2008 ορίστηκε το πλαίσιο δράσης, πρόκειται για ένα μέσο το οποίο είναι πλεονασματικό διότι δεν παρέχει προστιθέμενη αξία. Μιλά με γενικούς όρους και δυστυχώς δεν άλλαξαν τα νομοθετικά συστήματα των κρατών μελών. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για το οργανωμένο ε, έγκλημα με το αποτύπωμα της μαφίας. Τον Αύγουστο του 2010 Ρώτησα την Επιτροπή κατά πόσο γνωρίζει την οικονομική επίπτωση της δράσης της μαφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι στην Ιταλία αυτή η οικονομική επίπτωση ανέρχεται σε 135 δις ετησίως. Ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πόσο γνωρίζει αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής και μίλησε για την Καμόρα, την Τράγκετα, την Κόζα Νόστρα, όλες τις διακλαδώσεις δηλαδή της μαφίας. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αντιμεταπίσουμε επαρκώς. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν έχει σύνορα, δεν είναι ιταλικό πρόβλημα, δεν ε, περιορίζεται στην ιταλική επικράτεια. Εγώ μιλώ για τις ελλείψεις της χώρας μου, αλλά μπορώ να πω σε όλους ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα να εξαγάγουμε την ομοθεσία μας ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με ε, αποτύπωμα της μαφίας γι' αυτό. Από δικαστικής και πολιτικής πλευράς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ιταλικό, καθαρά αφορά την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αυστρία, για να, αναφέρω, να αναφερθώ σε ορισμένες μόνο χώρες. Και Εκεί έχουν ριζωθεί, έχει ριζωθεί η μαφία και αναλαμβάνει και δραστηριότητες συντονισμού. Πρόκειται για ένα ευφυές δίκτυο το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εκεί όπου υπάρχουν ευίωνοι οικονομικοί όροι για να μπορέσει να δράσει ατιμωρητή. Άρα εμείς οι Ευρωπαίοι βουλευτές. Εάν δεν ε, το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε ο καθημερινός αγώνας της Ιταλίας δεν θα είναι αποδοτικός εάν οι άλλες χώρες υφίστανται τις συνέπειες. Εάν μολυνθούν, γιατί πρόκειται για έναν ιό, ο οποίος μολύνει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα καρκίνωμα, μία νεοπλασία, η οποία όλο ένα και επεκτείνεται. Πρόκειται για την χειρότερη οικονομική και πολιτισμική εκδήλωση, πολιτισμική εκδήλωση θα μπορούσα να πω, της χώρας μου. Δυστυχώς οι ευρωπαϊκές αρχές υποτίμησαν το πρόβλημα. Κάθε χώρα το αντιμετώπισε ξεχωριστά αυτό το ζήτημα με βάση την νομοθεσία της. Όμως, όπως ανέκυψε από την ακρόαση της 29ης Μαρτίου, προέκυψαν ουσιώδη ζητήματα που αφορούν και την συνδρομή και συνεργασία των δικαστικών αρχών. Ο Ισαγγελέας Γκρατέρη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εμπειρογνώμων καταπολέμησης της Ντράγκετα ανά τον κόσμο, αναφέρθηκε σε ειδικά μέτρα και συγκεκριμένες δράσεις σε άλλες χώρες και είπε ότι θα πρέπει μέσα στα πλαίσια της Eurojust να είμαστε σίγουροι για αυτό το δίκτυο συνεργασίας και τις αιτήσει συνεργασίας. Η συνεργασία της Eurojust δεν αρκεί. Πολλές φορές μιλάμε για ε, δράση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κολομβία ή στο Βέλγιο, διότι υπάρχει καλή σχέση μεταξύ δικαστικών αρχών, διμερός, δηλαδή μεταξύ Ιταλίας και Κολομβίας ή Ιταλίας και Βελγίου. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτό. Θα πρέπει να πω ότι η Ευρώπη είναι πεπισμένη ότι το πρόβλημα της μαφίας αφορά ορισμένες χώρες αποκλειστικά, ιδιαίτερα την δική μου. Αυτή η συλλογιστική είναι λανθασμένη και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο είναι ριζωμένο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το να ακολουθούμε τακτική στρουθοκαμιλισμού στην Ιταλία ονομάζεται ομερτά, δηλαδή το δίκαιο της σιωπή. Και αυτό ενισχύει τη μαφία. Υπό αυτή την έννοια η εμπειρία της Ιταλίας θα πρέπει να αποτελέσει δίδαγμα για όλους. Λυπάμαι εάν τα λόγια μου φαίνονται κοινότοπα, αλλά εμείς έχουμε ζήσει στο πετσί μας αυτή την πραγματικότητα, την επίπτωση του οργανωμένου εγκλήματος. Γνωρίζουμε εκ πρώτης ότι θα πρέπει να έχουμε μία αποφασιστική πορεία καταπολέμησης και συνεργασία, δικαστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι εάν δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να είναι αμόλυντη από τις 27 χώρες, μόνο τότε θα μπορέσει να αντιδράσει. Δεν υπάρχουν σύνορα στο οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Δεν υπάρχουν γεωγραφικά σύνορα για τη μαφία. Το οργανωμένο έγκλημα δημιούργησε ένα δίκτυο συνένεσης με πολιτικές διεισδύσεις, διείσδυση στη νόμιμη οικονομία και στην δημόσια διοίκηση. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούν ενδοκοινοτικός και εξοκινοτικός οι χώρες. Υπάρχει η μαφία της Αλβανίας, της Νιγηρίας, της Ρωσίας, τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού. Έχουμε να κάνουμε με πραγματικές πολυεθνικές που δρούν μέσω της νόμιμης οικονομίας. Είναι εμβληματική η περίπτωση της ντράγκετα. Η ντράγκετα, τα έσοδα της ντράγκετα ισοδυναμούν με το ΑΕΠ έξι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οργανωμένο έγκλημα λοιπόν δρά διεθνικά και διασυνοριακά και έτσι θα πρέπει να ειδωθεί. Άρα δεν υπάρχουν σύνορα ενδοκινοτικός για το οργανωμένο έγκλημα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια ευρωπαϊκή δράση. Δυστυχώς όμως ενδοκινητικος υπάρχουν σύνορα. Η συνθήκη της δυνατότητας παρέχει νέες δυνατότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας και από την άποψη των οργάνων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, δύο συνοριακά. Europol, Eurojust, Όλαφ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Θα πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση. Βεβαίως πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο θα πρέπει να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις γιατί υπάρχει διαφορετικό σύνταγμα στα κράτη-μέλη. Πρόκειται όμως για ένα όργανο το οποίο θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνθήκες μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέμβουμε με βάση ένα κοινό πλαίσιο και θα πρέπει να κινηθούμε αμελητή προς αυτή την κατεύθυνση με βάση τις ευθύνες μας. Θα πρέπει να αρχίσουμε λέγοντας τι πρέπει να καταπολεμήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα σαφή ορισμό που να ισχύει, ισχύει για τα 27 κράτη-μέλη. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, πώς το ορίζουμε. διότι μιλάμε για προστιθέμενο πολλαπλασιαστικό ε, μέσο όρο συνδρομής, μάλλον μέσο όρο συνδρομής που θα δράσει πολλαπλασιαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τον χαρακτήρα της κάθε οργάνωσης, να δούμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για απειλές και για οργανωμένο έγκλημα και έτσι θα είμαστε σίγουροι για την σοβαρότητα. Άρα με βάση το 416α θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το αποτύπωμα της μαφίας με βάση συγκεκριμένες δικαστικές και ανακριτικές έρευνες. Μιλώ για την δυνατότητα παρέμβασης με φυλάκιση και με συλλήψεις δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης και θα πρέπει η Κομισιόν να υποβάλει μία πρόταση οδηγίας. Αυτό που έχει σημασία είναι η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και η συνεργασία δικαστικής αρρωγής και συνεργασίας. Αυτό είναι σημαντικό για να φτάσουμε σε μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορέσει να δράσει κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν μπορώ να σας ε, μιλήσω για τις μεμονωμένες προτάσεις, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Η εγκληματικές οργανώσεις είναι σε δράση να μπορέσουν να ριζωθούν και να πλήξουν χιλιάδες οικογένειες. Δυστυχώς οι πολιτικές ε, τάσεις δεν είναι αποτελεσματικές. Μιλάμε για την εκμετάλλευση και την κατάσχεση και ελπίζω η Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε την Κομισιόν έτσι ώστε να προβάλλει μια φιλόδοξη πρόταση. Θα πρέπει να εκριζωθεί το οργανωμένο έγκλημα και όλα του τα πλοκάμια από τον οικονομικό ιστό και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε δράση κατά της ανακύκλωσης του χρήματος για να μην μολυνθεί ολόκληρος ο οικονομικός ιστός και να υπάρχει διαφορά μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου. Επίσης, ασχολήθηκα με την υποστήριξη των θυμάτων και της οικογένειας του, τους. Πολλές φορές ε, τα θύματα, οι οικογένειες πρέπει να ζήσουν μια δραματική κατάσταση και πολλές φορές ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, το πρόβλημα στην ολότητά του επειδή στη χώρα μου έχουμε ζήσει αυτό το πρόβλημα της ε, μαφιόζικης τρομοκρατίας, θεωρώ ότι αυτά τα θύματα θα πρέπει να υποστηριχθούν. Πλήττονται από ένα σύστημα το οποίο προσπάθησε να γονατίσει όχι μόνο μία ολόκληρη χώρα, αλλά και να πλήξει τη δημοκρατία αυτού του κράτους. Ως προς τους μάρτυρες, πολλοί επιχειρηματίες άρχισαν να μιλούν κατά της μαφίας που τους εκβιάζει. Και θέλουμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ε, μάρτυρες. Δυστυχώς αυτό δεν ήρκεσε. Εγώ ελπίζω να υπάρξει καλύτερη προστασία όταν ένας ε, μάρτυρας υποστηριχθεί με 100.000 ευρώ μπορεί να πληρώσει τα χρέη του, αλλά ένας επιχειρηματίας δεν θα μπορέσει να ξαναργαστεί γιατί θα έχει γύρω του καμένη γη. Όταν λοιπόν ένας ε, επιχειρηματίας γίνεται δικαστικός μάρτυρας θα πρέπει να έχει προτιμησιακές οδούς για να μπορέσει να ξαναεργαστεί. Πολλά είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε τα δημόσια έσοδα να μην μπουν στις τσέπες της ε, μαφίας σε σχέση με το δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ο τύπος και ο πολίτης να μπορέσει να διαβουλεύεται και να βλέπει πού χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα online. Αυτό το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα του Κοινοβουλίου. και δεν μπορεί να μην μας ενδιαφέρει το συλλογικό συμφέρον. Θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να, φέρουν, να έχουν κώδικες συμπεριφοράς για να καταδικάζουν το οργανωμένο έγκλημα σε όλες τους, τους, τις εκφάνσεις. Το σημείο εκκίνησης είναι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόσκομα στο να υπάρξει δικαιοσύνη και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να έχω μεγάλη συνεισφορά των σκιωτών έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτή η έκθεση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άλλο δικαστή που σκοτώθηκε στην Ιταλία. Αυτός ο δικαστής έδειξε ότι θα πρέπει να αγαπούμε τη χώρα μας ακόμα και όταν δεν μας αρέσει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ο δικαστής αυτός ήταν ο Πάολο Μπορσελίνο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και επειδή μιλούσα ιδιαίτερα γρήγορα θα δώσω το Λόγω στον ε, ε, ισαγγελέα Νταλτέριο, ο οποίος ασχολήθηκε στη Νάπολη με την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων της μαφίας. Την περασμένη εβδομάδα μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθώ και με άλλους δικαστές που δουλεύουν στο συγκεκριμένο αυτό τομέα και καταγράψαμε την τρέχουσα κατάσταση με αυτούς τους δικαστές δύο ημέρες εντατικής εργασίας ε, σε μια ακρόαση που βελτίωσε κατά πολύ τις γνώσεις μας ε, επί του θέματος. Εγώ είχα προσκληθεί ως εμπειρογνώμων και ομολογώ ότι ως εμπειρογνώμων πολλές φορές έχω κάνει σφάλματα. Διδάσκομαι όμως από τα σφάλματά μου. Και θα έχω την ευκαιρία και μαζί σας να συζητήσω αυτά τα οποία έχω αποκομίσει από την εμπειρία μου από το 1992 όταν ο κύριος Φαλκόνη και ο κύριος Μπροσελίνο ε, δολοφονήθηκαν έχουμε διδαχθεί πολλά. Δημιουργήθηκε το Γραφείο εισαγγελία κατά της μαφίας και έγιναν πολλές έρευνες οι οποίες δεν είχαν πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έκτοτε έχουμε βελτιώσει κατά πολύ τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε κατά της μαφίας. Εγώ έχω ασχοληθεί με την κατάρτιση δικαστών εδώ και τα χρόνια και νομίζω ότι κάτι που μας βοηθάει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι ότι έχουμε τώρα εμπειρίες τις οποίες μπορούμε να ανταλλάσσουμε με άλλα κράτη-μέλη. Δημιουργήθηκε ε, γραφείο καταπολέμησης των δραστηριοτήτων ε, της μαφίας πριν από λίγα χρόνια στην πρώην ε, Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Ιουκοσλαβίας, στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε μια χώρα δηλαδή που επρόκειτο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δώσαμε τη δυνατότητα και εμείς με την εμπειρία μας στην Ιταλία να εκπαιδευθούν δικαστές στην ε, γειτονική χώρα. Ε, από τις εμπειρίες μας λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και άλλους καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο σχέδιο έκθεσης που σας παρουσίασε η κυρία Αλφάνο υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι καρπός αυτής της εμπειρίας. Υπάρχουν απειλές από τη μαφία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και η απειλή της μαφίας είναι συνεχής και έντονη. Έχουμε κάνει πολλέ προόδου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, όπω σα είπα, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα το ίδιο έχει κάνει προόδου. Ε, δεν υπήρχαν ποτέ σύνορα για οργανώσει τύπου μαφία και πριν από την πτώση του τείχου του Βερολίνου και μετά υπάρχει διεθνή συνεργασία και η μαφία αλλάζει συνεχώ πρόσωπο με τα ίδια αποτελέσματα. Προσπαθούν να υπονομεύσουν θεσμού, να υπονομεύσουν την κοινωνία και την δημοκρατία. αντικαταστάθηκαν 180 ε, τοπικοί εκπρόσωποι από το 2000 και υπάρχει ε, και το διάταγμα 267 σχετικά με τα μέτρα κατά της μαφίας και λόγω ε, των της εισχώρησης της μαφίας σε τοπικές αρχές μετακινήθηκαν από τη θέση τους 180 ε, τοπικοί εκπρόσωποι. Παρότι ε, είχαν ε, χάσει το αξίωμά τους, εξελέγησαν εκ νέου και χρειάστηκε και πάλι να μετακινηθούν από τη θέση τους. Η Καμόρα, η Ντράγκετα από την Καλαβρία και Ε, ε, είναι οργανώσεις τις οποίες ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και υπάρχουν δεσμοί με τη μαφία σε άλλες χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μάθει ότι η Ιταλική μαφία ε, προσπάθησε ε, να ε, μπει στη συμφωνία και στη σύμβαση για την ανοικοδόμηση του Ground Zero, στο χώρο δηλαδή όπου είχαν γίνει οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη το 2001, συνεργαζόμενοι με την τοπική μαφία. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 φάνηκε ότι εξαφανιζόταν η Κόζα Νόστρα, διαχωριζόταν σε πολλά κομμάτια και μπήκε στην παρανομία εγκαταλείποντας τις εγκληματικές και δολοφονικές επιθέσεις κατά των δικαστών, αλλά έσπασε σε πολλά τμήματα Προσπαθώντα να αντιμετωπίσει την καταπολέμηση της μαφίας από τι ιταλικέ αρχές. Επειδή υπάρχουν όλε αυτέ οι προσπάθειε με τους μάρτυρε που υποστηρίζονται, με τους πληροφοριοδότες, η Κόζα Νόστρα και η μαφία έχουν διαχωριστεί σε πολλά κομμάτια, σε πολλού μικρούς πυρήνε και οι ερευνητέ δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη σαφή ιεραρχία της μαφίας που υπήρχε στο παρελθόν. Στο παρελθόν υπήρχε μια ξεκάθαρη ιεραρχία την οποία μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς. Και η Ντράγκετα τώρα δεν βασίζεται μόνο σε οικογενειακούς ε, δεσμούς. Είναι πιο εξειδικευμένο το δίκτυο της Ντράγκετα. Λειτουργεί και στην Καλαβρία και στη Λομβαρδία τώρα είναι αποκεντρωμένοι πλέον και οι πυρήνες της δουλεύουν αυτόνομα. Και η Καμόρα συνεχίζει να είναι ε, κατακαιρματισμένη και δεν έχει συνενωθεί με άλλες οργανώσεις Και είναι πιο δύσκολο να βρούμε πληροφορίες για μέλη της Καμόρα τώρα, ενώ στο παρελθόν υπήρχε μια ιεροτελεστία για να γίνει κανείς μέλος της Καμόρα και ήταν πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε την ιεραρχία της οργάνωσης. Ο Τομάσο Πουσέτο είπε ότι δεν υπάρχει μαφία, υπάρχει η Κόζα Νόστρα. Η Κόζα Νόστρα δεν θα είχε γίνει μαφία αν δεν είχε συμμαχήσει, όπως το έχει ήδη κάνει με σημαντικούς τομείς της κοινωνίας των πολιτών, με τον οικονομικό τομέα, με τον τομέα της δημόσιας διοίκησης, με τις επιχειρήσεις, με πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και μετά από χρόνια έρευνας διαπιστώνουμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Και παρότι έχουμε επιτύχει πολλά από πλευράς του δικαστικού τομέα, δεν έχουμε μειώσει τον κίνδυνο από την απειλή αυτών των οργανώσεων τύπου μαφίας. Η μαφία επικρατεί όταν η κοινωνία των πολιτών είναι αδύναμη, όταν δεν υπάρχει αξιοκρατία και όταν η κοινωνία των πολιτών αποδέχεται το νόμο της ζούγκλας, αποδέχεται τις σχέσεις και τις ε, δωροδοκίες και όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ε, κάνουν πραγματικά τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν. Θυμάμαι τον Τζοβάνι Παλκόνη που μιλούσε για ένα ε, μαφιόζο που τον ρώτησε ο δικαστής τι είναι η μαφία και είπε σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχει μια κενή θέση για έναν εισαγγελέα και να έχουμε ένα εισαγγελέα ο οποίος είναι άξιος και έχει δουλέψει καλά και ένας άλλος υποψήφιος ο οποίος έχει σχέσεις ε, με τη μαφία. Ε, θα είναι προτιμότερος αυτός ο οποίος δεν θα έχει δουλέψει καλά, αυτός ο οποίος δεν θα έχει αναλάβει δράση. Γιατί αυτό αναμένει η μαφία από τους εισαγγελείς, να μην αναλάβουν μέτρα. Εμείς έχουμε περάσει στην αντίθετη κατάσταση, δηλαδή έχουμε αναλάβει ενεργό δράση, έχουμε λάβει μέτρα κατά της μαφίας και προσπαθούμε να έχουμε και συνταγματικές εγγύησεις. Στη χώρα μας έχουμε υιοθετήσει νόμους για να αντιμετωπίσουμε την μαφία. Έχουμε πολύ αποτελεσματική νομοθεσία τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει τη διάρκεια των ποινών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δίμευσης της περιουσίας μελών της μαφίας. Ελέγχουμε αυτούς οι οποίοι κερδίζουν δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις, εξετάζουμε τα υποστηρικτικά έγγραφα σε ε, προκηρύξεις διαγωνισμών, προσπαθούμε να σταματήσουμε το ξέπλυμα χρημάτων, δεν θέλουμε οι καρποί της παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας της μαφίας να εισραίουν εκ νέου ως νόμιμα έσοδα στην ε, κανονική οικονομία και όταν αναλαμβάνει κάποιος ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει να υποβάλει μια δήλωση που να εγγυάται την ακαιρεότητά του χωρίς παράλληλα να μειώνουμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε να έχουμε και υψηλότερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και καταπολέμηση της μαφίας. Αυτοί που δουλεύουν στο δικαστικό και αστυνομικό τομέα θέλουμε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και θέλουμε και η νομοθεσία μας να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε γιατί είναι πολύ έξυπνη η μαφία. Παρισφρεί στην κοινωνία των πολιτών, παρισφρεί στην αγορά. Χρησιμοποιεί ε, κάποια πρόσωπα που είναι η εικόνα της προς τα έξω, είναι κάποια πρόσωπα βιτρίνα και καταφέρνει να μπαίνει ε, στις επιχειρήσεις, ε, στην κοινωνία των πολιτών, παραβιάζοντας την νομοθεσία, παραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία, παραδείγματο χάρη. Δεν συνεργάζονται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όσοι έχουν καταδικαστεί από την Τράγκετα υποχρεώνονται ε, να καταβάλουν αποζημίωση 10 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια λόγω της μη ανάπτυξης της περιοχής που οφείλεται στην Τράγκετα. Είναι μέτρα αποτρεπτικά αυτά, είναι μέτρα τα οποία δείχνουν ότι όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και οι δικαστές πρέπει να εγγυώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προστατεύουν τα συμφέροντα αυτών που έχουν θυγεί από τη μαφία και η πολιτεία πρέπει να λάβει δράση κατά της μαφίας μέσω του εισαγγελέα της δίκη κατά της Μαφία. Ξέρω ότι δεν έχω ε, πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και θα προσπαθήσω να φτάσω σε κάποια συμπεράσματα. Συμφωνώ με τι βασικές προτάσει που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. ιδίω θα ήθελα να αφαιρθώ στα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ε, ενεργειών είναι ένας ε, τομέας που πρέπει περαιτέρω να αναπτύξουμε, ο τομέας της προστασίας των θυμάτων. Τα θύματα θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο το απόλυτο δικαίωμα σε οικονομική υποστήριξη Ε, και τα θύματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ε, στην ερευνητική διαδικασία, να μπορούν ε, να θέτουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν στη δικαστική διαδικασία υποβοηθώντας την, το ρόλο των δικαστών. Θύματα που έχουν θυγεί λόγω της μαφίας θα πρέπει να συμμετέχουν στη δικαστική διαδικασία. Ξέρω βέβαια ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να σας δώσω τόσες λεπτομέρειες. Θα είχα πολλές λεπτομέρειες να σας δώσω γιατί η μαφία είναι ένα πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη πολύ συγκεκριμένα. Το οργανωμένο έγκλημα έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα και διαπράττονται πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα τα οποία είναι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να σκεφτούμε τις απάτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας λάβουμε υπόψη την Καμόρα πώς έχει δράσει στο τομέα της διατροφής. Η Κόζα Νόστρα, τι έκανε στο βιομηχανικό τομέα, η Ντράγκετα, τι έκανε στον ενεργειακό τομέα και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν εμπλακεί στην αγορά εργασίας και στον οικονομικό ιστό με παράνομες δραστηριότητες χωρίς να τηρήσουν τους κανόνες της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει και τι κάνει. Κάνει αρκετά. Εμείς οι δικαστές που καταπολεμούμε τη μαφία βλέπουμε ότι δίνονται πολλές οθήσεις σε πολλούς ε, τομείς για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να προσαρμόσουν την εσωτερική ένωμη τάξη στη, στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο με βάση την κύρωση των συμβάσεων όπως εκείνη στις 29 Μαΐου 2000 για την δικαστική αρρωγή και την ε, συνεργασία των δικαστικών αρχών. διότι η δικαστική συνδρομή χορηγείται με βάση την πρώτη δικαστική αρχή που ζήτησε τη συνδρομή. Άρα, το πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί σχετίζεται με τον τομέα της δικαστικής αρρωγής ή συνδρομής. Αρκεί να δείτε ε, την ευαίσθητη συνεργασία με βάση τις αποφάσεις πλαίσιο του 2003, 5 και 6 σε σχέση με την ε, κατάσχεση αγαθών που είναι απότοκα ε, ιδεχθών οικονομικών πράξεων. Λίγες είναι οι χώρες ε, που ανταποκρίνονται τάχιστα και που μπορούν να ανταποκριθούν με σπουδή και που έχουν κατανοήσει ότι όταν πρόκειται για, βασικά, για τέτοια ε, ιδεχθή εγκλήματα θα πρέπει να δράσουν άμεσα. Δεν χρειάζεται εξ νόβο να εισαγάγουμε στοιχεία. Ελπίζω οι κοινέ ερευνητικές αρχές να μπορέσουν να δράσουν και να συνεργαστούν. Δυνάμει της απόφασης πλαίσιο της 13ης Ιουνίου 2002 για να μπορέσουν να δράσουν και η Eurojust και η Europol. Η Eurojust μπορεί να ε, μας δώσει πολλές οδηγίες για να μπορέσουμε να δράσουμε. Οι ερευνητικές αρχές επιτρέπουν να μπορέσουμε να δράσουμε μέσα στα πλαίσια των μεμονωμένων κρατών μελών. Μέσα στα πλαίσια της αμοιβαία δικαστικής σύνδρομης ευχαριστούμε τον ε, εισαγγελέα Αλτέριο Ναι, θα λάβετε το λόγο κι εσείς, απλώς πρέπει να δώσω το λόγο στην Επίτροπη πρώτα. Έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε και τόσο πολύ χρόνο. Ο κύριος Τινέ έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ εκπροσωπώ το Γενικό Διευθυντή για τι εσωτερικέ Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρχικά θα ήθελα να σα πω ότι όσον αφορά την έκθεση που τέθηκε υπόψη μα, χαιρετίζουμε σε γενικές γραμμές του στόχους της έκθεσης και υποστηρίζουμε ορισμένες από τις ενέργειες που περιέχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια οπωσδήποτε στιάστηκαν στο οργανωμένο έγκλημα ως σημαντικό φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμήσουμε με σκοπό να δημιουργηθεί ένας χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην Ευρώπη. Συνεπώς χαιρετίζουμε αυτή την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως συνομοθέτες. Όσον αφορά τώρα ορισμένα σημεία τα οποία αναφέρει η έκθεση και ανέφερε ο κύριος Αλφάνο, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε την έκκληση που απευθύνει το Κοινοβούλιο στις πολιτικές δυνάμεις, ώστε να υπάρξουν περισσότεροι πόροι ε, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και για να διευκρινιστεί ότι υπάρχει πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, δυστυχώς, συμφωνούμε τις ανησυχίες που διατύπωσαν ορισμένοι ομιλητέ σήμερα σχετικά με την αυξανόμενη διείσδυση των εγκληματικών οργανώσεων σε διάφορους τομείς, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στον κόσμο της οικονομίας ε, και των τραπεζών, κυρίως όσον αφορά την ομοθεσία Όσον αφορά την ποινικοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος, έχουμε μια έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί στα πλαίσια της υπάρχουσας απόφασης πλαισίου τον ερχόμενο χρόνο και καταρχήν το Μάιο του 2012 θα δημοσιευθεί και η έκθεση αυτή θα είναι η βάση για πιθανές μελλοντικές προτάσεις από την Επιτροπή. Θα ήθελα εδώ να επενθυμίσω ότι ήδη όταν εγκρίθηκε αυτή η σημαντική έκθεση η Επιτροπή είχε διατυπώσει επιφυλάξεις σχετικά με το ότι το έγγραφο δεν προσέθεται μεγάλη προστιθέμενη αξία σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία και υποστηρίχθηκε σε αυτή τη σκέψη η Επιτροπή από την Ιταλία και τη Γαλλία. Ένα θέμα χρόνου εδώ. Η έκθεση προτείνει ή μάλλον καλεί την ε, Επιτροπή να παρουσιάσει μία πρόταση μέχρι το τέλος ε, του έτους, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατόν. Διότι αν είχαμε αποφασίσει να ενεργήσουμε σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογή, θα έπρεπε να είχε γίνει μία μελέτη επιπτώσεων και αυτό ε, θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο. Συμφωνούμε όμως απόλυτα με την προτινόμενη πρόταση για την κατάσχεση και την ανάκτηση των προσφυγικών στοιχείων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα πρώτα απ' όλα με την προσπάθεια συλλογής των προϊόντων του εγκλήματος και σκοπεύουμε φέτος να παρουσιάσουμε μια φιλόδοξη πρόταση για την κατάσχεση και την ανάκτηση των περιφερειακών στοιχείων και θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο όσον αφορά το ουσιαστικό δίκαιο και την αμοιβαία ε, αναγνώριση. Θα συνεργαστούμε από αυτού με τις υπηρεσίες ε, της ε, Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα δικαιοσύνης. Αυτό θα αποτελέσει μέρος ενός πακέτου για την προστασία της οικονομίας κατά της διείσδυση των εγκληματικών οργανώσεων. Επίσης θα περιλαμβάνονται μέτρα πολέμηση απάτης στα σχέδια μια στρατηγικής ε, της Όλαφ και καταπολέμηση της διαφθοράς. Όσον αφορά τώρα το κοινωνικό θέμα, θα ήθελα να σας πω ότι στο παρόν στάδιο αναλύουμε, εξετάζουμε πολλές, πολλές διατάξεις αυτής της αναθεώρησης και η κοινωνική διάσταση περιλαμβάνεται στην ανάλυση, αλλά η αξιολόγηση επιπτώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι πρόωρο το στάδιο για να σας πούμε κατά πόσον ε, θα υπάρξει πρόβλεψη στην πρόταση της Επιτροπής αυτής της διάστασης. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε συντομία σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Το θέμα της προστασίας των θυμάτων, το οποίο επίσης υπογραμμίζεται και αναφέρθηκε πολύ και στην ε, έκθεση και στην ακρόαση, εδώ σύντομα θα κάνει μια νομική πρόταση η Επιτροπή η οποία στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται ότι περιλαμβάνει την προστασία των πληροφοριοδοτών και των θυμάτων. Αυτό βεβαίως είναι της ευθύνης της κυρίας Ρέντινγκ. Τώρα, σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες, χαιρετίζουμε την πρόταση της έκθεσης να δημιουργηθεί μια επιτροπή σε αυτό το κοινοβούλιο για τις ε, εγκληματικές οργανώσεις μαφιόζικες, νομίζουμε ο τύπου μαφίας δηλαδή, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και υποστηρίζουμε και τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να βελτιωθούν οι γνώσεις για το οργανωμένο έγκλημα, κυρίως τις επιπτώσεις του εγκλήματος αυτού στην κοινωνία. Ως προς τη μελέτη που προτείνεται στην Επιτροπή να αναλάβει θα ήθελα να σας κάνω την εξή πρόταση. Δεδομένου ότι πολλές από τις πληροφορίες που θα πρέπει να διατεθούν για να έχει νόημα αυτή η μελέτη είναι πληροφορίες από τις διοκτικές αρχές και καλό θα ήταν να συμμετάσχει σε αυτή τη μελέτη και η Europol ώστε να έχουμε ορισμένα στοιχεία που ένας εξωτερικός ερευνητής δεν θα μπορούσε ίσως να βρει. Επίσης υποστηρίζουμε τις ενέργειες που έχουν σχέση με την Eurojust και την αμοιβή αναγνώριση. Επίσης, όσον αφορά την εκπαίδευση του δικαστικού σώματος και των αστυνομικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια, μια προτεραιότητα, όπως είδατε στα οικονομικά μας προγράμματα στην Επιτροπή, τόσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της δικαστικής δικαιοσύνης. Ποινικής δικαιοσύνης. Συμφωνώ επίσης ότι το θέμα της διαφάνειας του δημοσίου τομέα είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το παράδειγμα της ε, Ιταλίας, αλλά το γεγονός ότι τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι αναγνεύσιμα και να τα παρακολουθούμε, είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στη δική μας την αντίληψη, η οποία θα παρουσιαστεί ε, στην ε, προσεχή στρατηγική καταπολέμηση της απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα όπου συμφωνούμε απόλυτα με το σχέδιο έκθεσης είναι το θέμα καταπολέμησης διαφθοράς. Αυτό είναι ειλικρινά ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε πολλές μελέτες. Το Ευρωβαρόμετρο άλλωστε βρίσκεται στο επίκεντρο των ε, προβληματισμών των πολιτών 78% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρσι είπαν ότι κατά τη γνώμη τους η διαφθορά ήταν μείζον πρόβλημα στη χώρα τους και η Επιτροπή σκοπεύει στα πλαίσια του πακέτου για την προστασία των οικονομιών να προτείνει μέσα καταπολέμησης της διαφθοράς όπως ένα μηχανισμό αξιολόγησης της προόδου καταπολέμησης της απάτης στα κράτη-μέλη. Συνεπώς μία νέα έκθεση για ε, την ε, διαφθορά. Και θα περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα όπως μια εφαρμοστική έκθεση για την απόφαση ε, πλαίσιο για τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα και έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τον μηχανισμό αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βεβαίω, τα μέτρα κατά του ξεπλήματος του χρήματος είναι πολύ σημαντικά, όπως και η πρόθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της καλλιέργειας της νομιμότητας. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, επειδή δεν υπάρχει χρόνος θα σταματήσω εδώ. Ήδη αυτή η έκθεση είναι πολύ περιεκτική και πιθανό θα θέλαμε να υπογραμμιστεί και το θέμα ε, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Δεδομένου ότι οι διοκτικές αρχές αναφέρουν όλο και περισσότερο ότι μέσω του διαδικτύου το διαδίκτυο ε, διευκολύνει όλες τις συμβατικές μορφές εγκλήματος και επιτρέπει, είναι ένα όργανο επικοινωνίας. Γι' αυτό θα έπρεπε να το παρακολουθούμε καλύτερα και οι εθνικές στρατηγικές κατά του οργανωμένου εγκλήματος στρέφονται προς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πιστεύουμε. Επίσης μιλήσαμε πολύ για την αξιολόγηση της απειλής. Εδώ θα έπρεπε ίσως να υπογραμμίσουμε το ρόλο της Europol ώστε να κάνει στρατηγικές αξιολογήσεις ε, ε, απειλών που θα αποτελέσουν τη βάση της ανάλυσης των άλλων θεσμικών οργάνων και βρίσκονται και στη βάση ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ολοκληρώνω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στην Προεδρία, στον Δ. Πέτερ Στάουμπερ από την Ουγγρική Προεδρία. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω διότι με καλέσατε ως εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω αυτά που κάνουμε εμείς για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ την κυρία Αλφάνο για την έκθεσή της. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα πλήρης περιλαμβάνει εξαιρετικές προτάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα αγώνα ο οποίος θα διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τίθεται και προτεραιότητες για την καταπολέμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην παρουσίασή μου θα σας αναφέρω τις βασικές προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας κατά τους έξι μήνες της Προεδρίας μας. Θα ήθελα εισαγωγικά να αναφέρω κάτι που τόνισε ο Ούγγρος Υπουργός Εσωτερικών τον Ιανουάριο, Σάντον Πίντερ, είπε ποιο είναι το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας και είπε ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος έγινε μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας για διάφορους λόγους. Ε, κύριος λόγος είναι ότι το πρόβλημα αυτό είναι διεθνές, μας επηρεάζει όλους και υπάρχουν και αντίστοιχες εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο. Άλλος ένας λόγος είναι ότι έχουμε δει ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα θέμα εσωτερικής ασφάλειας που μέχρι τώρα δεν έχει τύχει της πρέπουσας σημασίας. Τρίτον, βλέπουμε ότι μετά την κρίση υπάρχει μια αλλαγή στις στρατηγικές τις οποίες εφαρμόζει το οργανωμένο έγκλημα και πρέπει να αποδώσουμε σημασία ακριβώς σε αυτή την αλλαγή από πλευράς οργανωμένου εγκλήματος. Τα μέτρα τα οποία εμείς έχουμε λάβει είναι τα εξής. Στις 20 Ιανουαρίου έγινε στο Γκέντελε μία άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών και ήταν παρόν και ο κύριος Λόπεθ, ο πρόεδρος σας, και έκανε και μία παρουσίαση σε, αυτό το, αυτή τη συνεδρίαση. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ήταν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έλαβε το λόγο ο διευθυντής της Europol, ο γενικός γραμματέας της Interpol και το κέντρο ΣΕΚΙ που έχει τα γραφεία του στη Βουδαπέστη ε, παραβρέθηκε μέσω του διευθυντού του. Αναφέρθηκαν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές, οι πρόσφατες τάσεις στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και όχι στατικό, αλλάζει τις στρατηγικές του και ε, μετά την ε, οικονομική κρίση έχει τροποποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του. Το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί τις αγορές, η αγορά όμως έχει αλλάξει και οι οργανωμένες ομάδες του εγκλήματος αναζητούν ευκαιρίες και νέες ευκαιρίες στις ε, νέες αγορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανακατανομή των ε, αγορών που είναι διαθέσιμες για το οργανωμένο έγκλημα. Οι Υπουργοί συζήτησαν τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος συμφώνησαν ότι πρέπει ε, να αυξήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε διεθνές επίπεδο καθώς και με οργανισμούς όπως η Europol, η Interpol και οργανισμοί όπως ε, το κέντρο ΣΕΚΙ που έχει έδρα στη Βουδαπέστη. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα. Οι Υπουργοί επίσης συζήτησαν και κάτι άλλο το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση είπαν ότι ε, η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων είναι ένα βασικό σημείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εθνικές στρατηγικές ε, σχετικά με την ε, δίμευση των χρημάτων που είναι απόρρια δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθείται μια διατομεακή προσέγγιση που έχει αποδώσει αποτελέσματα και τέτοιου είδους μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αναφέρεται και στην έκθεση της κυρίας Αλφάνο αυτό. Μια άλλη δραστηριότητα της Ουγγρικής Προεδρίας είναι ότι συνεχίζουμε το έργο της Βελγικής Προεδρίας Η Βελγική Προεδρία πέρυσι τον Νοέμβριο κατέληξε ε, σε κάποια ε, συμπεράσματα για ένα μηχανισμό και έναν κύκλο πολιτικών που καλύπτει διετής και τετραετής περιόδους και καθορίζει προτεραιότητες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εμείς στην Ουγγρική Προεδρία ολοκληρώνουμε ένα τμήμα, μια περίοδο αυτού του μηχανισμού. Η Europol είχε προετοιμάσει την έκθεση ΟΚΤΑ για την αξιολόγηση των απειλών από το οργανωμένο έγκλημα και με βάση την έκθεση αυτή εμείς ετοιμάζουμε τα συμπεράσματα για το Συμβούλιο Υπουργών του Ιουνίου που θα θέσει τις προτεραιότητες για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό θα αφορά και δράσεις της ε, αστυνομίας και ε, δράσεις συνεργασίας. Έχουμε αρχίσει λοιπόν αυτή η διαδικασία προετοιμασίας του Συμβουλίου του Ιουνίου. Μία άλλη δράση είναι ότι υπάρχει μια ομάδα που θα είναι τμήμα της ε, Επιτροπής Ασφάλειας της ΚΟΖΗ Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Φινλανδία, Πολωνία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Europol συνεισφέρουν στις εργασίες αυτές των οποίων ηγείται η Ουγγαρία και αυτή η ομάδα θα ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο. Στο εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφεται η πολυτομεακή προσέγγιση την οποία σας προανέφερα. Θέλουμε να καταγράψουμε τις ορθές πρακτικές και βέλτιστες πρακτικές σε αυτό τον τομέα, ούτως ώστε με αυτό το εγχειρίδιο να ενημερώνονται οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θέλουμε να καταγράψουμε όλες τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες έχουμε εντοπίσει και να το δώσουμε αυτό το εγχειρίδιο στα κράτη-μέλη για να έχουν χρήσιμα παραδείγματα. Προχωρούμε αρκετά καλά με το εγχειρίδιο αυτό και ελπίζουμε ότι θα το έχουμε ολοκληρώσει μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ιουνίου. Θα συνεδριάσει άλλη μια φορά η ομάδα που ασχολείται με την κατάρτιση του εγχειριδίου και μετά τη συνεδρίαση αυτή θα ολοκληρωθεί και το εγχειρίδιο και θα ολοκληρώσει την εργασία της αυτή η ομάδα εργασίας με το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα μείνει όμως ως αποτέλεσμα και κληροδότημα για το μέλλον αυτό το εγχειρίδιο. θα συζητήσουμε στην ομάδα εργασίας και το πώς θα είναι δυνατόν να ενημερώνεται αυτό το εγχειρίδιο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δώσατε το λόγο να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση. Συγχαίρω την κυρία Αλφάνο για την εξαιρετική της έκθεση και βεβαίως θα είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα αρχίζει η συζήτηση. Έχουν Anchis, Borsellino e bronze. Ο κύριος Ιακολίνο ε, μπορεί να δώσει τα λεπτά του στον κύριο Κροτσέτα. Ο κύριος Κροτσέτα για τρία λεπτά. Εκτιμώ την έκθεση και την εισήγηση της κυρίας Αλφάνο καθώς και όσα ελέγχθησαν από τον κύριο Αλτέριο και την Κομισιόν. Στις 15 Ιουλίου 2009 έγραψα στον πρόεδρο Μπούζεκ για να ε, μελετηθεί συστηματικά αυτό το φαινόμενο. Και Δυστυχώς αυτή η μελέτη δεν διενεργήθηκε, αποτελεί ε, υπόσχεση η οποία δεν ε, εκπληρώθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα με βάση την εμπειρία βουλευτών που προέρχονται από τις διάφορες χώρες. Εγώ στις 15 Ιουλίου του 2011 πάλι θα γράψω στο Μπούζεκ γιατί αυτή η Επιτροπή κατά της Μαφίας δεν έχει συσταθεί παρόλο που το έχω ζητήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ένα λάθος. Δεν πρέπει το πρόβλημα της μαφίας να απορρέει από το γεγονός ότι η Ιταλία απασχόλησε την Ευρώπη. Τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Δηλαδή, η μαφία πια δράσε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει και σήμερα υπάρχουν νέες μαφίες όχι μόνο στην ε, Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για μαφία δεν μιλάμε μόνο για την Τράγκετα, την Κόζα Νόστρα, την Καμόρα. Πρέπει να μιλήσουμε για την ε, ε, Αλβανία, Βουλγαρία, Κίνα, Ρωσία, Νιγηρία, την Κολομβία και το ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι εθνικές μαφίες. Ποιο είναι το πρόβλημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν μιλάμε για οικονομικό έργο θα πρέπει να μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, αλλά αυτό αποτελεί μεγάλη υποκρισία, διότι όλοι χρησιμοποιούν το μοντέλο Κόζα Νόστρα, που είναι η μόνη μορφή οργανωμένου εγκλήματος που δεν νικήθηκε από κανέναν. Ποιο είναι το μοντέλο είναι η σχέση μεταξύ οικονομικού και είναι διασύνδεση μεταξύ οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού τομέα. Και σας δίνω αυτό το παράδειγμα γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου του 2003 ως δήμαρχος είχα αρχίσει να καταπολεμώ τη μαφία και οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο μαφιόζους. Ο ένας ήταν Σικελός και ο άλλος ε, Λιθουανός. Ε, συζητούσαν για το πώς θα με εξοντώσουν. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2003 θα συνέβαινε κάτι το πολύ σημαντικό που θα άλλαζε τα δεδομένα στη Σικελία και Λιθουανία. Τότε είχε αποφασιστεί η εισδοχή της Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έγινε λόγος για, από πλευράς προεδρίας για οργανωμένο έγκλημα. Αλλά αυτό είναι καθαρά υποκριτικό, διότι όλα πάντα προσυμφωνούνται. Θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τη μαφία με τη Eurojust, τη Europol και θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταπολεμούμε την ε, παράνομη μετανάστευση. Εάν οι δικαστικές αποφάσεις σημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες Κύριε Κοσέτα, πρέπει να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα. Δεν υπάρχει καμία αμοιβαιότητα σε σχέση με θέματα δικαστικής αρρωγής. Πάντα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, διότι οι Γάλλοι με ρωτούν, μα υπάρχει ακόμα αυτή η απειλή. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν κατανοούν τίποτα για τη μαφία. Θέλουμε λοιπόν να ε, προωθήσουμε αυτή τη μελέτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να συσταθεί μια ερευνητική επιτροπή για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο κύριος Γιακολίνο. Μ' αρέσει να είμαι απίθαρχος και τα κατάφερα πολύ καλά στη ζωή μου ακριβώς επειδή είμαι απίθαρχος. Μιλάει εκτός μικροφώνου ο κύριος Γιακολίνου και δεν τον ακούμε. Νομίζω ότι γίνονται πολλές εκτιμήσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δική σας πρόταση. Δεν υπάρχει ε, καμία αμφιβολία ότι το οργανωμένο έγκλημα επιβάλλει μία δομή ανταπάντησης. Δηλαδή η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα υπό το φως της συνθήκης της Λισαβόνας και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που ορίζει τη μέθοδο συνεργασίας με τρίτες χώρες για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να δούμε το καρτέλ της Κολομβίας, ε, την Ιγυρία με την εμπορία ανθρώπων και ούτω καθεξής, καθώς και την παράνομη χρήση ευρωπαϊκών πόρων. Όπως υπογραμμίστηκε και από την προηγούμενη παρέμβαση, υπάρχουν ορισμένοι πυλώνες που προβλέπονται στην ε, Ιταλική νομοθεσία. Αυτή η εμπροστοφυλακή δεν δημιουργήθηκε έξι μήνες πριν. Πρόκειται για μια νομοθεσία το, του τέλους της δεκαετίας του 70 και που θα πρέπει να θεωρηθεί μοντέλο αναφοράς γιατί θα πρέπει να ανακτήσουμε τα χρήματα τα οποία δόθησαν αχρεωστήτως στις ε, αρχές του εγκλήματος. Και η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει καλύτερα και τους ε, μηχανισμούς κατάσχεσης. Και έχουμε και το 49 το 41α, το οποίο αφορά τις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Αγαπητή Σόνια, βεβαίως ορισμένα θέματα θα πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, υπάρχει και η διεφθαρμένη πολιτική, αλλά και μια πολιτική που αντιτάσσεται στη μαφία. και στο 8 και 9 μιλάς για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της μαφίας. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα θύματα. Τι θα γίνει με την Ειδική Ερευνητική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ Μιλήσαμε για την της, εμπροστοφυλακή της ε, Ιταλίας. Υπάρχουν και συγκεκριμένες δομές πολέμησης της απάτης. Θα πρέπει να δούμε τι θα, κάνει και, τι θα κάνουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός εδώ. Εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα ελευθεροτυπία όπως νομίζουμε. Θα πρέπει να δούμε τι ποιοτικά άλματα μπορούμε να κάνουμε. Μην ξεχνάμε και το άρθρο 27 του Συντάγματος που αναφέρεται στην πολιτική γειτονίας. Γιατί να μην προβλέψουμε και μέτρα πρόληψης που αναγνωρίζουμε από την ομοθεσία μας. Από την μας. να δούμε τι θα γίνει και με τη σύμβαση του 2000. Οπωσδήποτε θα πρέπει να αναφερθούμε και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία ολισθαίνει και προς τα αλλού. Πρέπει να εξευρωπαίσουμε την έννοια αυτή και τα μέτρα. Και τελειώνω πριν από το συνάδελφο Κροτσέτ. έχω λίγο περισσότερο χρόνο. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 3 Μαΐου. Σε, στο πολυσχηδές αυτό θέμα που μας απασχολεί. Εγώ θεωρώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 3 Μαΐου. Αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα άλλο πλαίσιο, τότε θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα έγγραφο που να συμβαδίζει με τις πραγματικές μας ανάγκες. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Γιάνσκης. Άγκης. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα με το οποίο ασχολείστε είναι ένα από τα σημαντικότερα. Στην αρχή εξηγήσατε ότι αυτή η έκθεση ήταν προσωπικό θέμα για σας. Εδώ έχουμε ορισμένε συγγένειε, αν θέλετε, διότι και για μένα είναι προσωπικό θέμα. Όχι μόνο δηλαδή ένα ζήτημα πολιτικής ή ένα ζήτημα έρευνας, αλλά είναι το οργανωμένο έγκλημα και η διασύνδεση με τις ε, πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι πολύ σημαντική τα, τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, είδαμε πολλές περιπτώσεις διαφθοράς με βάση ε, το οργανωμένο έγκλημα, το ρωσικό ή το ρωσόφωνο οργανωμένο έγκλημα και ε, σε σχέση με εγκληματικούς κύκλους δυστυχώς σε υψηλά κυβερνητικά επίπεδα. Για μένα που έζησα σε μια κομμουνιστική χώρα το θέμα του ρωσικού ή ρωσόφωνο, όπως λέμε, οργανωμένου εγκλήματος, είναι κάτι το πολύ σημαντικό και έχει σχέση με τη διαφθορά. Και είναι και προσωπικό μου θέμα, το βλέπω προσωπικά. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το, τα δικά σας θέματα. Σκεφτήκα ότι ίσως σε κάποια ομάδα εργασίας ή σε κάποιο άλλο πλαίσιο, δεν ξέρω ποιο θα ήταν το καταλληλότερο, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον για μας να αναλύσουμε συστηματικά τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των εγκλημάτων της μαφίας και των εγκλημάτων που γίνονται από ρωσικές οργανώσεις, ρωσόφωνες εγκληματικές οργανώσεις. Το θέμα είναι ότι θα ήταν καλό να δούμε τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι η μαφία κατέκτησε ορισμένε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό σίγουρα συμβαίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται σε πολλά σημεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και στους, στα θεσμικά όργανα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως και στο Κοινοβούλιο, δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε, δηλαδή τι μέσα διαθέτουμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα ε, ή μάλλον την καταπολέμηση της διείσδυσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φυσικά, αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό σοβαρά. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ τώρα σε ένα θέμα μεθοδολογίας δεν είναι σαφής η μεθοδολογία, ε, δεν είναι σαφής η διάκριση. Μιλάμε ε, αδιακρίτως μερικές φορές για το οργανωμένο έγκλημα ή για τη μαφία. Δεν είναι το ίδιο. Η μαφία είναι μια μορφή ε, οργανωμένου εγκλήματος. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε εδώ και 150 χρόνια και περισσότερο στην Ιταλία. Όταν όμως μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα λέμε μαφιόζικου τύπου. Και αυτό περιλαμβάνεται ήδη ε, στο σύνταγμά μας από το 1982. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ε, τη διαφορά που υπάρχει και χρειάζεται ένα αιώνα για την αντιληφθούμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Πρόκειται για δύο πολύ επικίνδυνες πραγματικότητες και όπως λες στην έκθεσή σου με σαφέστατο τρόπο ε, όταν αναφέρεσαι σε οργανισμούς που ε, έχουν μεγάλες επιπτώσεις κυρίως στον οικονομικό τομέα. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η μαφία. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εργανομένη εγκληματικότητα μαφιόζικου τύπου είναι κάτι το διαφορετικό. Και πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση για να υιοθετήσουμε μέτρα Άλλωστε το συζητήσαμε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπενθύμησε ορισμένα σημεία, ορισμένα πράγματα τα οποία έγιναν στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και από την Επιτροπή μας. Ίσως επειδή υπάρχει αυτή η ιδιομορφία στα πλαίσια της Επιτροπής μας, είμαστε πολύ από τη Σικελία και ζήσαμε και υποστήκαμε τις συνέπειες αυτής της πραγματικότητας. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι μέσω αυτής της έκθεσης να κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε μία ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Διότι είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην Ιταλία. Όταν μιλούσαμε ε, για τη μαφία ως ένα μεσογειακό ή μάλλον πρόβλημα του Νότου θα έλεγα, η, η συνείδηση άλλαξε ε, στην Ιταλία και χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να αλλάξει η αντίληψη της ιδιομορφίας του φαινομένου της μαφίας. Αν λοιπόν και στην Ευρώπη επιθυμούμε να αναλάβουμε κοινά μέτρα και αποτελεσματικά, ουσιαστικό είναι να υπάρξει αυτή η συνειδητοποίηση όσον αφορά την ιδιομορφία αυτών των οργανώσεων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που συνδέονται μεταξύ τους φυσικά. Ε, το ένα φαινόμενο είναι η συνέπεια του άλλου, παρόλα αυτά όμως είναι δύο φαινόμενα διαφορετικά, ευδιάκριτα. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μπρόνς. Σας ευχαριστώ. Η, συνθήκη, η έκθεση λέει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, προσφέρει νέες δυνατότητες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση, τουλάχιστον στο παρελθόν, διευκόλυνε την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος λόγω της εξάλληψης των συνόρων ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και κεφαλαίου. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεται διακίνηση ανθρωπίνων ε, ανθρώπων όταν δεν υπάρχουν σύνορα στον ε, χώρο ε, του, του Σέγγεν. Όπως επίσης και ελεύθερη διακίνηση νομίμων προϊόντων και παρανόμων αντικειμένων όπως όπλων και ναρκωτικών. Και η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου αφήνει και τη δυνατότητα για το ξέπλυμα χρήματος. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερη ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με την έκθεση. Το μήνυμα το οποίο παίρνω είναι ότι η δημιουργία εθνικών συνόρων εκ νέου θα δημιουργούσε ε, την ευκαιρία για ένα χτύπημα κατά κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτοί που είναι υπέρ της ενοποίησης της Ευρώπης συνεχώς μιλούν για τις απειλές και είναι πραγματικές οι απειλές από το οργανωμένο έγκλημα για να αυξήσουμε την δυνατότητα ε, αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος ε, υπάρχουν μέτρα όπως το Europol, η Interpol και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Έχω ένα πρόσθετο ερώτημα. Αναφέρθηκε το θέμα της διείσδυσης της μαφίας ε, στον επιχειρηματικό νόμο νόμιμο κόσμο. Πάντοτε υπάρχει συνέχεια της δραστηριότητας της μαφίας όταν έχουν διεισδύσει σε αυτές τις επιχειρήσεις ή υπάρχουν στοιχεία ότι το προσωπικό της μαφίας ε, που ενδεχομένως θέλει να ξεφύγει από την οργάνωση αυτή ε, ε, χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αυτή για να φύγει από την παράνομη δραστηριότητα και μετά δρούν σχετικά νόμιμα στον επιχειρηματικό κόσμο. Δεν θα ήθελα τέλος τα σχετικά αρνητικά μου σχόλια να ε, ε, θεωρηθούν ε, σχόλιο κατά της εξαιρετικής έκθεσης της κυρίας Αλφάνο και θα ήθελα να επενέσω και το θάρρος της. Allora, ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Και θα δώσω το λόγο στον ε, εισαγγελέα για τα δικά του συμπεράσματα και στη συνέχεια θα εξαγώ και εγώ τα δικά μου συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε ένα τεχνικό ερώτημα σχετικά με την εμπειρία των δικαστών ε, για την καταπολέμηση της μαφίας. Και ο κύριος Μπρόνς έκανε μια σχετική ερώτηση για τα μέσα που χρησιμοποιούν αυτοί που βρίσκονται εκτός μαφίας για να έρθουν σε επαφή με τη μαφία και να επωφεληθούν από τις δραστηριότητε της μαφίας. υπάρχει μια συναλλαγή μεταξύ μαφίας πολιτικής και επιχειρήσεων. Αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Η περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε αφορά τις δραστηριότητε μαφίας, ε, καμόρα, ντράγκετα και ούτω καθεξής μέσα στα πλαίσια των προεκλογικών εκστρατείων και υπόσχεσεων σε εκδήλωση ενδιαφέροντος σε διαγωνισμούς. Άρα πολλές φορές γίνονται αναθέσεις σε επιχειρηματίες και αναδόχους παράνομα με βάση συγκεκριμένα, συγκεκριμένο αντίτιμο βεβαίως. Και έτσι εξασφαλίζεται και η κοινωνική ειρήνη μέσα στα πλαίσια των επιχειρήσεων με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Στο παρελθόν είχαμε να κάνουμε με τη μαφία καταρχήν τον επιχειρηματικό κόσμο και την πολιτική, δηλαδή τους εκπροσώπους των πολιτικών αρχών και των θεσμικών οργάνων. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται, θα χρειαζόταν να παρέμβω πολύ περισσότερο με βάση τα δεδομένα. Θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι και αυτές οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Υπό την έννοια ότι αντί να, να έρθουμε σε επαφή με, τη, με τις επιχειρήσεις, οι μαφίες το κάνουν αυτό. Πολλές φορές οι σχέσεις έχουν, είναι εξασφαλισμένες ως προς την διασύνδεση μαφιόζων και επιχειρηματικού κόσμου. Εμείς θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στον Φραντσέσκο Καμπανέλα που είναι συνεργάτης και που ανήκει στην Κόζα Νόστρα της Σικελίας και ομολόγησε την ευθύνη του. Ήταν επιχειρηματίας και διευθυντής ε, ενός ε, υποκαταστήματος, τραπεζικού υποκαταστήματος. Ανακύκλωνε το χρήμα της ε, Κόζα ε, Νόστρα και ήταν και δημοτικό σύμβουλο στο Παλέρμο. Ερχόταν σε επαφή λοιπόν με τους επιχειρηματίες και τους τοπικούς πολιτικούς. Αν λοιπόν ρωτήσουμε τι σχέσεις υπάρχουν, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μία. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι η μαφία ανακυκλώνεται διότι στο εσωτερικό της υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα για να μπορέσει να ελέγχει την επικράτεια και τον κοινωνικό ιστό. Ευχαριστούμε τον Ισαγγελέα Νταλτέριο. Θα ήθελα να πω το εξής. Εάν συμφωνείτε ως προς τις προθεσμίες θα μπορούσαμε να ειδωθούμε στις 19 ε, το απόγευμα κατά τις 2.30 για να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα υποβληθούν οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, ως προς τις παρατηρήσεις του κυρίου ε, Κροσέτα, θυμάμαι πότε το ζήτησες αυτό από τον ε, πρόεδρο Μπούζεκ, γιατί και εγώ προσυπέγραψα και έστειλα ένα γράμμα υποστήριξης στον πρόεδρο Μπούζεκ για να τονίσω το γεγονός ότι χρειάζεται μία επιτροπή διενέργειας έρευνας κατά των δραστηριοτήτων της μαφίας, όπου θα πρέπει να συμμετέχουν οι κυβερνητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές και ούτω καθεξής. Ε, δηλαδή, ε, όσοι δρούν και γνωρίζουν το θέμα. Για μένα αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Ο κύριος Αλτέριο αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ως προς τον κύριο Γιακολίνο θα ήθελα να πω, όπως είπα και πριν, ότι η νομοθεσία κατά της ε, μαφίας αποτελεί έναν απόσπαστο στοιχείο της δραστηριότητές μας και θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γιατί η μαφία είναι ένα φαινόμενο που εξάγεται, ένα εξαγώγημο προϊόν. Σε σχέση με τη σκληρή φυλάκιση, το άρθρο 41α, εγώ μπαίνω στη θέση συναδέλφων που βρίσκονται μακριά από μας. Εκεί όπου η μαφία θεωρείται ένα θέμα folklore δηλαδή λαϊκού χρώματος. Δηλαδή ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα μία αυστριακή συνάδελφος μας είπε ότι σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, θεωρείται ένα θέμα ε, καθαρά τοπικού ε, ένα θέμα που έχει τοπικό χαρακτήρα, ένα θέμα φολκλόρ αν θέλετε να εκφραστώ έτσι. Και Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ισχύει και για τις 27 χώρες. Αυτό που τόνισε και ο Ισαγγελέας Νταλτέριο. Γιατί θα πρέπει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σφαγή τη ε, Duisburg Τότε οι Καλαβριανοί είπαν ότι θα πρέπει στο εστιατόριο Νταμπρούνο να διερευνηθεί η κατάσταση εκεί δηλαδή που έγινε η μεγάλη σφαγή και να δούμε κατά πόσο οι αρχές αρνούμενες αυτή την απαγωγή δεν επέτρεψαν στις δικαστικές αρχές να προβούν προς συγκεκριμένε έρευνες. Όταν μιλάμε λοιπόν για συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, μιλάμε ακριβώς γι' αυτό. Άρα συμφωνώ ότι θα πρέπει να ε, ανταποκριθούμε και στη σκληρή φυλακή, δηλαδή στο άρθρο 41α της εσωτερικής μας ένομης τάξης έτσι ώστε ο καταδικαστής να μην μπορεί να δίνει εντολές από τη φυλακή ή να έχει διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Αναφερθήκατε και στον τύπο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μιλάμε για ελεύθερο τύπο, ο οποίος δεν υπόκειται σε εκφοβισμούς γιατί μην ξεχνάτε ότι οκτώ δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τη μαφία, έχουν δολοφονηθεί από τη μαφία. Και κάνοντας αυτή τη διαπίστωση βλέπουμε ότι οκτώ ε, δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην Ιταλία, αλλά αυτό αφορά και την Ισπανία και την Κολομβία και ούτω καθεξής και ο τελευταίος δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε ήταν ο ίδιος μου πατέρας. Η συνάδελφος Άγκης για τη ρωσική μαφία υπάρχει η έκθεση του δόκτωρος Σκαρπινάτο του Ισαγγελέα που θεωρεί ότι το 40% των ιδιωτικών επιχειρήσεων και το 60% των δημοσίων και το 85% των ε, τραπεζών της Ρωσίας υπόκεινται επιρροή από το οργανωμένο έγκλημα. Και οι μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις την χάνουν διαχείρισης του ρωσικού εγκλήματος. Επίσης δωροδοκούνται βουλευτές. Οι 450 βουλευτές της Δούμα χρησιμοποιούν 15.000 βοηθούς, εκ των οποίων πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στα πλαίσια ε, μαφιόζικων δραστηριοτήτων. Αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο στοιχείο των υποδομών του καπιταλισμού, του γεωπολιτικού καπιταλισμού. Πρόκειται για τον ίδιο τρόπο δράσης, έχουμε να κάνουμε το ίδιο modus agendi που ισχύει ανά τον κόσμο. Και ελπίζουμε να συσταθεί μια κοινοβουλευτική επιτροπή κατά πολέμησης της μαφίας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που μας προείπατε. Μπορσελίνο. Και εγώ μίλησα για αυτή τη διάκριση, έτσι ώστε να γνωρίζουμε κατά πόσο πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα ή για τη μαφία. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,5 χρόνο πριν πρότεινε το UCBN και εγώ τότε το απέρριψα κατέβαλα μεγάλες προσπάθειες για να γίνει κατανοητό ότι δεν πρέπει να μιλάμε για έγκλημα, διότι το έγκλημα καθε αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα γενικότερα. Αλλιώς μιλάμε για υπόκοσμο. Όπως τόνισες και εσύ, θα πρέπει να μιλάμε ε, για οργανωμένο έγκλημα με, αποτύπωμα, με το αποτύπωμα της μαφίας. Και εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις. Εμείς με αυτή την έκθεση αποτελεί κόλαφο για τους συναδέλφους, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν συνειδητοποιήσει την εμβέλεια του ζητήματος. Εμείς προσπαθήσαμε να φτάσουμε ιεραρχικά σε αυτό το συμπέρασμα, βαθμιαία μάλλον, διότι μέχρι πρότινος ε, δεν γινόταν λόγος για οργανωμένο έγκλημα στο Κοινοβούλιο. Σήμερα μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα με το αποτύπωμα της μαφίας έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην μπορούν να γυρίσουν προς τα πίσω. Να μιλάνε για μία απτή πραγματικότητα, μία πραγματικότητα που μας αφορά όλους αδιακρίτως. Δεν υπάρχει μία χώρα που να μην συμμετέχει. Και καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε μέχρι πρότινος, δηλαδή να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πρέπει να το κάνει υπέρ των πολιτών. Όταν η Σουηδική Προεδρία και ο επικεφαλής των αστυνομικών αρχών μου είπε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες, θα πρέπει να πούμε ότι και στη Σουηδία υπάρχει η μαφία. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Καλύτερα λοιπόν να δείξουμε ότι έχουμε υποτιμήσει το πρόβλημα παρά να, πούμε, να κάνουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να προσποιούμαστε δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τα στοιχεία από εσάς έτσι ώστε να δείξουμε ότι αναγνωρίζουμε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους καταπολεμώντας το οργανωμένο έγκλημα. Σας ευχαριστώ. Noi. ευχαριστούμε. Eh, ευχαριστούμε την κυρία Αλφάνο. Εργαστήκατε πολύ καλά και ευχαριστούμε και τον Ισαγγελέα Νταλτέριο που καταπολεμά τη μαφία και οι τροπολογίες θα υποβληθούν, λέει ο πρόεδρος και διακόπτη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όπως μας είπε η κυρία Αλφάνο. γιατί πρόκειται για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Siamo un po' in ritardo. Έχουμε καθυστερήσει κάπου. If you please, we're following, following to... Παρακαλώ, περνάμε τώρα στο σημείο 11. Η εσωτερική στρατηγική ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η συγγήτρια είναι η κυρία Ρίτα Μπορσελίνο. Δεν είναι εδώ. Όχι, εντάξει. Έρχεται, έρχεται come ¿Eh? το έγγραφο εργασία. Έχουμε το πολύ 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Διότι ως συνήθως έχουμε καθυστερήσει. Λόγω της φορτωμένης ημερήσιας διάταξης. Έχουμε λοιπόν 30 λεπτά για ανταλλαγή απόψεων ε, πάνω σε ένα έγγραφο εργασία το οποίο έχει υποβληθεί από την εισηγήτριά μας την κυρία Ρίτα Μπορσελίνο. Θα μας μιλήσει η κυρία Μπορσελίνο και κατόπιν θα μπορέσουν να μιλήσουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους, αλλά για λόγους υγείας χρειάστηκε να αναβάλουμε την παρουσίαση αυτού του εγγράφου και έγινε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ο όρος ασφάλεια η λέξη ασφάλεια αυτές τις τελευταίες μέρες ε, μας δείχνει ότι δεν σημαίνει τίποτα αν δεν συνοδεύεται από τη λέξη αλληλεγγύη. Κανένα μέσο ασφάλειας δεν θα λειτουργήσει εάν στην Ευρώπη είμαστε μοναχικός καβαλάρης. Κυρίως θα έλεγα ότι θα έχουμε και αρνητικές επιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν κάθε πλεονέκτημα να συνεργάζεται κανείς με άλλους, θα πρέπει να βασιστούμε ε, στα μέσα που διαθέτουν οι συνθήκες. Τα δύο έγγραφα εργασίας που παρουσιάζω αναφέρονται στα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Το ζητούμενο δεν είναι να επινοήσουμε νέες μεθόδους, νέα εργαλεία, εάν δεν κάνουμε πρώτα απολογισμό των όσων υπάρχουν. Βλέπετε λοιπόν στο έγγραφό μου από πού ξεκινάμε και τι διαθέτουμε. Ε, στο τομέα των προτάσεων αυτό θα γίνει μέρος της έκθεσης που θα παρουσιάσω τον Ιούνιο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η εξέλιξη της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα είναι καρπός τελευταίων εξελίξεων, δεδομένου ότι αυτό το θέμα δεν είχε περιληφθεί από τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, εφόσον ήταν θέμα εθνικής κυριαρχίας. Αλλά το πρώτο παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών ήταν η συνθήκη του Σέγγεν, το οποίο θεωρήθηκε ως δευτερεύον μέτρο ε, στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτός ο μηχανισμός επέτρεψε να ενοποιηθεί η πολιτική των θεωρήσεων, να δημιουργηθεί δικαστική συνεργασία, αστυνομική συνεργασία και τα κράτη-μέλη αυτού του χώρου, του Σέγγεν, ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν και την εσωτερική ασφάλεια ε, στα πλαίσια του Σέγγεν. Και σε αυτά τα πλαίσια υπήρξε κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα, κατόπιν ακολούθησαν οι συνθήκες ε, του Μάστρικ, του Άμστερνταμ και όλα αυτά έγιναν η κινητήριος δύναμη ε, ενός κράτους ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας έγινε ο δεύτερος στόχος. Ε, δεν, λοιπόν, δεν πρέπει λοιπόν να εκπλησόμεθα από το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας εφόσον χρειάστηκαν πάνω από 30 χρόνια για να ελοπιθεί η κοινή αγορά πρέπει να καθορίσουμε κοινέ πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις στον τομέα, τον πολιτιστικό, τον δικαστικό, τον πολιτικό ε, που αντικατοπτρίζουν αιώνε εθνική πολιτική. Η διαδικασία λοιπόν είναι μια διαδικασία ανοικοδόμηση. και το πρόγραμμα Τάμπερ του 1999 έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ανέδειξε αυτές τις διαφορές αλλά πρέπει επίσης να υπάρχει συντονισμός στα πλαίσια της καταπολέμησης των ναρκωτικών και των ανθρώπων κυρίως. Στις 11 Σεπτεμβρίου επίσης, η 11η Σεπτεμβρίου μάλλον, κατέδειξε την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας στρατηγικής ασφάλειας πέραν των άλλων πολιτικών της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία των κρατών μελών. Το ζητούμενο ήταν να βρεθούν στρατηγικές κανόνες που να αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια όλα τα κράτη-μέλη υποστήριξαν τη σημαντική μεταφορά αρμοδιοτήτων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια και, στο, και στη συνταγματική συνθήκη και στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Επίση, Εξαλήφθησαν ορισμένοι δισταγμοί όσον αφορά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά υπάρχει ακόμα αντίδραση όσον αφορά ε, τα στρατιωτικά θέματα και την εξωτερική ασφάλεια. Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερική ή την εξωτερική ασφάλεια. Αυτό όμω ε, μπορεί να καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την ενσωμάτωση μέτρων που βασίζονται σε μια δυναμική και σε ένα δικαστικό πλαίσιο που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μας υποχρεώνει όμως να καταφεύγουμε σε διάφορα μέσα. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης μεταξύ άλλων έδωσε επιπλέον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Αλλά απομένουν τρεις γκρίζες ζώνες που περιπλέκουν τον καθορισμό μιας κοινή στρατηγικής. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για την αλληλενέργεια μεταξύ εσωτερική και εξωτερική ασφάλειας. Η εσωτερική ασφάλεια και το ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο και μεταξύ των θεσμών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στην πρώτη περίπτωση, σχέση μεταξύ αρμοδιοτήτων της Ένωση στον τομέα της άμεσης ασφάλειας και την αρμοδιότητα στην εσωτερική ασφάλεια, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ένα ειδικό καθεστώς βάσει του οποίου όταν πρόκειται για ασφάλεια και άμυνα δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν νομοθετικές πράξεις και οι διεθνείς συμφωνίες δεν μπορούν να έχουν την ίδια δεσμευτική ισχύ όπως οι συμφωνίες που βασίζονται στις κανονικές αρμοδιότητες της Ένωσης, στον αστυνομικό και δικαστικό τομέα, το ποινικό δίκαιο. Και στα πλαίσια των κανονικών αρμοδιοτήτων, η συνθήκη προβλέπει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ενημερώνεται πλήρω σε αυτό το χρόνο στη διάρκεια διαπραγματεύσεων και κυρίως έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να εγκρίνει την συμφωνία. Σε αυτά τα πλαίσια οι διεθνείς συμφωνίες θεωρούνται ω η εξωτερική ε, επέκταση των συμφωνιών τη Ένωση και θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την αρχή τη Ευρωπαϊκή Πολιτική που ισχύει μετανάστευση, προστασία δεδομένων και ούτω καθεξής. Δηλαδή οι εσωτερικές ε, αρμοδιότητες ορίζουν τις εξωτερικές και όχι το αντίστροφο, όπως βλέπουμε σε ορισμένα έγγραφα του Συμβουλίου. Και υπό το φως αυτών των στοιχείων είναι ουσιαστικό να επιμείνουμε επί της συνεργασίας με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Με την Επιτροπή μας. Υπάρχει και μια άλλη γκρίζα ζώνη η εσωτερική ασφάλεια των χωρών αλλά και η εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας η πολιτική εσωτερική ασφάλειας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πλήρης ευρωπαϊκή πολιτική όπου ισχύουν οι αρχές που εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η άμεση εφαρμογή των κανόνων και η περιοχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια της δημόσιας ασφάλειας πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ο Ευρωπαίος νομοθέτης να σέβεται τα κριτήρια της επικουρικότητας και της αναλογικότητας για να αποφύγει προσφυγές στη δικαιοσύνη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το ίδιο το πρόγραμμα της Στοχόλμης διευκρινίζει ορισμένους στόχους και εξηγεί ποιο θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμικών οργάνων τη και των κρατών μελών. Το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει την απειλή στην εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης δημιούργησε ένα μηχανισμό όπου συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη με τη βοήθεια των οργανισμών Ευρωπόλ, Φροτέξ κυρίως και κόζι, άρθρο 71 των συνθηκών, αυτή, αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει να εστιάζονται τα μέτρα που είναι απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ εθνικών διοικήσεων είτε για να πραγματοποιηθούν στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και από αυτού θα υποβάλω προτάσεις στην έκθεση του Ιουνίου επειδή τα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπουν να πράξουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η έκταση της απειλής και θα θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στο όνομα καταπολέμησης αυτής της απειλής. Τρίτη γκρίζα ζώνη, σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενισχυτικό το γεγονό ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο αγνόησαν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώ και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στον ορισμό τη ε, στρατηγική ασφάλεια. Θεωρώ αδιανόητο αυτό το γεγονό. Αλλά τα βασικά έγγραφα τα οποία υιοθετήθηκαν αγνοούν παντελώ την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δημιουργούσε απορία και πριν από την άνοιξη ισχύω τη συνθήκη Λισαβόνα. Αλλά είναι ακόμα περισσότερο απορία άξιον το γεγονό ότι ένα χρόνο μετά από την ισχύ αυτή τη συνθήκη, πώ μπορούμε να περιμένουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μεταφράσει σε νομοθεσία ορισμένα στοιχεία τη στιγμή που δεν έχει ενημερωθεί πέραν από εκείνες που βρίσκει το Κοινοβούλιο μόνο μέσα από τον τύπο και θα αγωνιστεί το Κοινοβούλιο για να αναλάβει το ρόλο του. Απλά και μόνο αναφέρθηκα εγώ σήμερα στην υφιστάμενη κατάσταση. Αργότερα οι συνάδελφοι θα πρέπει να μας πούν τι πιστεύουν. Θα συναντήσω τους συνεισηγητές και όλους όσοι ενδιαφέρονται να ε, διατυπώσουν την άποψή τους. Αναφέρομαι στους δικαστές, για παράδειγμα. Δεν ζητήθηκε η γνώμη του. Αναφέρομαι στους υπεύθυνους ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρομαι στα εθνικά κοινοβούλια, στην Ευρωπόλ, την Eurojust, την Frontex κυρίω. Και άλλωστε υποφελούμε τη παρουσία τη επιτροπή για να τη απευθύνω ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στη βάση τη στρατηγική της ασφάλειας. Στο άρθρο 5 γίνεται λόγο για αύξηση ε, Τη δυνατότητα αντιμετώπιση της κρίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε επίσης για αξιολόγηση της απειλή. Έχω την εντύπωση ότι αν αφήσουμε αυτά στα κράτη-μέλη θα αυξηθεί η δυνατότητα αντίδρασης. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα βλέπουμε ότι η έκθεση παρουσιαστεί τον Ιούνιο και θα πρέπει όμως να γίνει και ένα ε, σεμινάριο των Εθνικών Κοινοβουλίων το Σεπτέμβριο. Αυτό το σεμινάριο του Σεπτεμβρίου των Εθνικών Κοινοβουλίων θα είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε το ρόλο που θα παίξουν αυτά τα κοινοβούλια κυρίω από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ελπίζω να υπήρξε αρκετά γρήγορη. Μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε όμως σχετικά αρχίσει και έχουμε να καλύψουμε κι άλλο ένα θέμα. Ο κύριος Νούνες Ντεαλμέιδα από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μπροσελίνο. Ε, καταρχήν θέλω να πω ότι η ενοποίηση ε, της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας από την Επιτροπή παρουσιάζει τις 21 δράσεις που θεωρεί προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, ε, αυτό είναι ένα έγγραφο που επικεντρώνεται στην ουσία περισσότερο και όχι στη θεσμική πραγματικότητα. Σαφώς και δεν είχαμε την πρόθεση να αμφισβητήσουμε τον νέο ρόλο του Κοινοβουλίου βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Απλώ αναφέρουμε τι δράσει που θεωρεί προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία με τα χαρά συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο για τον καθορισμό αυτής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων. Και με χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις ε, του Κοινοβουλίου για τους πέντε στόχους ε, και τις 41 ε, δράσεις που αναφέρουμε. Εγώ θα κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Έχουμε εντοπίσει πέντε βασικούς στόχους, τους οποίους μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία στην πράξη για την εσωτερική ασφάλεια. Για κάθε στόχο υπάρχουν κάποιες μετρήσιμες δράσεις. Δεν είναι πλήρη ο κατάλογο. Υπάρχουν πολλά τα οποία γίνονται και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο στόχο είναι η παρενόχληση των διεθνών δικτύων εγκληματικότητα. Μιλάμε για το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μετασχηματιστεί και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο βεληνικές. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία χάνει η οικονομία, χάνει η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Προσπαθούν ε, αυτά τα κυκλώματα να, να ζητούν τομείς της κοινωνίας όπου έχουν τη δυνατότητα να παρισφρήσουν. Ε, να διευκολύνουμε την, ε, το δικαστικό τομέα στην ερεύνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προβλέπονται δράσεις κατά της των μονάδων οργανωμένου εγκλήματος στην κοινωνία, καθώς και κατάσχεση των εσόδων από το παράνομο έγκλημα. Θέλουμε να δώσουμε νέα ορμή και να περάσουμε σε μια νέα αντιμετώπιση πέραν της παραδοσιακής πρακτικής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και μέσω της διοικητικής προσέγγισης ε, που θέλουμε να την κάνουμε πάρα πολύ αποτελεσματική σε περίοδο οικονομικής ε, δυσκολίας. Δεύτερος στόχος ε, να αποτρέψουμε την τρομοκρατία και την στρατολόγηση τρομοκρατών. Συνεχίζει να αυξάνεται η απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας και δεν θα πρέπει εμείς να χαλαρώσουμε την προσοχή μας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα απαραίτητα μέσα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε όλους τους τομείς της ασφάλειας. Πολλές σημαντικές δράσεις έχουν δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 100 μελών, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και άλλους εταίρους καταπολέμηση της χρήσης του διαδικτύου από τους ε, ε, τρομοκράτες, καταπολέμηση της ρίζοσπαστικοποίησης, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ρίζοσπαστικοποίησης, η ανακοίνωση της Επιτροπής μιλά για εταιρική σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που θα αυξάνει την επίγνωση αυτών των θέματων για την αύξηση των ριζοσπαστικών τάσεων. Ε, τρίτος στόχος, καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναπτύσσεται ταχύτατα και οι συνέπειες είναι ε, τραγικές για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις ε, και αποτελεί και απειλή για τις κρίσιμες υποδομές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί και να ερευνά το θέμα του, κυβερ... του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο μέσω ενός ειδικού κέντρου. Τα κράτη-μέλη και ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να διευκολύνουν την προστασία των πολιτών, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι πολίτε να προστατεύονται και να αναφέρουν περιστατικά εγκλήματο στον κυβερνοχώρο. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των πολιτών, για να αποφεύγεται η προτροπή προ τρομοκρατία. Τέταρτος στόχος, αύξηση της ασφάλειας μέσω της διαχείρισης των συνόρων. Πολύ συχνά τα ίδια άτομα είναι υπεύθυνα για την ε, διακίνηση ναρκωτικών και για τη διακίνηση ατόμων μέσω των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θέλει λοιπόν ε, παράλληλα να διαχειριστεί και του στόχου καταπολέμησης τη εγκλήματο ε, και του στόχου καταπολέμησης τη τρομοκρατία. και μέχρι τη θέση σε ισχύ τη ε, συνθήκης τη Λισαβόνας υπήρχε ένα τεχνητό διαχωρισμό στα σύνορα όσον αφορά τι απειλέ που τίθενται από άτομα και απειλέ που τίθενται από εμπορεύματα όπω τα ναρκωτικά ακόμη και αν οι ομάδε που διέπρεταν αυτά τα εγκλήματα ήταν οι ίδιε. Η ανακοίνωση τη Επιτροπή προτείνει τώρα μεθόδου για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, αυξάνοντας ε, το συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων οργάνων στα σύνορα. Ο στόχο υπαριθμών 5, για τον οποίο έχει υποβάλει και την ερώτησή της ε, η κυρία Μπορσελίνο, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένας στόχος για να αυξήσουμε την ε, δυνατότητά μας για αντιμετώπιση όλων των κρίσεων και ανθρωπογενών κρίσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, δημιουργία ε, μια αξιολόγησης κινδύνων, ε, στην οποία δεν θα ε, εμπεριέχονται καθόλου κίνδυνοι και παράλληλα έχουμε το στόχο να έχουμε μια πιο αποτελεσματική πολιτική ανταπόκρισης στις καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πρότεινε η κυρία Μπορσελίνο, θέλει να αποτυπώσει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, να αποτυπωθούν οι ανθρωπογενείς κίνδυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε καλύτερα την πολιτική μας. Αυτό θα αποτελέσει άλλο ένα βήμα για να οριμάσει ο ρόλος της πολιτικής, στο τομέα της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να παρέμβει σε δραστηριότητες επιβολής ε, του νόμου. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών με την πιθανή ε, υποστήριξη της Europol. Αυτό το οποίο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να υπάρχει είναι ε, μια δυνατότητα αξιολόγησης κινδύνων για τη δημιουργία πολιτικών για να βελτιώσουμε την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και της δημιουργίας δικτύων μεταξύ των εθνικών φορέων. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα τραγικά περισσότερο από ό,τι προσδοκούσατε από μένα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο σύντομο. Ήταν δύο σελίδούλε που θεώρησα σκόπιμο να σα διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και θα περιμένω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Δερμέιντα, αλλά σα υπενθυμίζω, λέει ο πρόεδρο, ότι μέχρι τι 12.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη συνεδρίασή μα. Μηπω θέλει το λόγο η Ουγγρική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Μπορσελίνο και θα ήθελα να πω ότι εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας χαιρετίζουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης ελπίζοντας ότι θα υιοθετηθεί εγκαίρως μέσα στις τακτές προθεσμίες. Θα είμαι σύντομος. Ήθελα μόνο να τοποθετηθώ επάνω σε ορισμένα σημεία. Και μεταξύ άλλων θα ήθελα να πω το εξή. Η Ουγγρική Προεδρία διατηρεί τις επαφές της με το Κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Μπούζεκ πριν από λίγο καιρό. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόοδο που έχει επιτελεστεί σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να γίνουν σεβαστά για προσχώρηση στο Σέγγεν. Αυτή την πρωτοβουλία την αναλάβανε με μετά από αίτηση του Κοινοβουλίου. Μιλώντας τώρα για διαφάνεια. Αυτό είναι προφανές και στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Μόλις άκουσε η Προεδρία να γίνεται λόγος για αυτό το σχέδιο έκθεσης της κ. Βουρσελίνο προσωπικά θέλησε να τη συναντήσω και στην αρχή Φεβρουαρίου της είπα ότι ήμασταν στη διάθεσή της για να τη βοηθήσουμε σε αυτό το εγχείρημα που είχε αναλάβει. Απλά σας επαναλάβω τι είχε γίνει και επαναλαμβάνω την προσφορά μας. Επίσης, ε, ανέφερα ότι η πρόεδρος της Κόζη, η κυρία Μπέρτα, ήταν διατεθειμένη να εμφανιστεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όποτε θελήσετε, ώστε η Επιτροπή σας να ενημερωθεί σχετικά με τις δραστηριότητες της Κόζη. Και αυτή την προσφορά μας την προτείνω και πάλι. Είμαστε έτοιμοι να έλθουμε κοντά σας, να σας δούμε και να σας ενημερώσουμε για τα όσα γίνονται στα πλαίσια ε, της Κόζη. Είμαι και αντιπρόεδρος αυτής της Επιτροπής, το οποίο σημαίνει ότι η Κόζη εκπροσωπείται εδώ από μένα. Θα ήθελα να κάνω και άλλη μια παρατήρηση. ότι εάν δείτε το άρθρο 72 της συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι αναφέρεται η δημόσια τάξη και η εσωτερική ασφάλεια ε, που ορίζονται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν άλλαξε τον ορισμό και οι κύριες δραστηριότητες της ΚΟΖΗ έχουν ως αντικείμενο την συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο και το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε αυτό το τομέα. Όπως ήδη είπα, είμαστε διατεθειμένοι να παρουσιάσουμε έναν απολογισμό της κατάστασης εδώ όταν το επιθυμείτε. Φυσικά, αυτά δεν ε, αμφισβητούν την αρμοδιότητα του συνομοθέτη που έχει το Κοινοβούλιο. Αλλά υπενθυμίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι μέχρι την 1η 12 2014 το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία στον τομέα της συνεργασίας των αστυνομικών δυνάμεων. Βεβαίως, η κάθε δραστηριότητα πρέπει να σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και το δικαστήριο δεν θα μπορεί να αποφανθεί επί των θεμάτων αυτών. Τελευταία παρατήρηση. Το Νοέμβριο 2010 η Επιτροπή είχε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για την υλοποίηση των στρατηγικών εσωτερικής ασφάλειας. Εκείνη την εποχή το Συμβούλιο είχε χαιρετήσει αυτή την έκθεση στις 24 Φεβρουαρίου και αυτό είναι σαφέστατο στα συμπεράσματα και η έκθεση για την εσωτερική ασφάλεια θα σταλεί στο Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του χρόνου και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας. Αυτά ήθελα να σας πω σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και για μία ακόμη φορά σας εύχομαι καλή τύχη στη συνέχεια των δραστηριοτήτων σας, κυρίως για την έγκριση της έκθεσης. Και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε την, τις υπηρεσίες μας. Για τους επόμενους ομιλητές παρακαλώ, όχι πάνω από 1,5 λεπτό, για να αφήσουμε λίγο χρόνο και για το τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης για σήμερα το πρωί. Κυρία Χάνκης, έχετε το λόγο πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν τα γνώριζα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Προσελίνο για την όλη συνεργασία. Είμαι σε δύσκολη θέση και δεν ξέρω τι να κάνω. Ω σκιώδης εισηγήτρια για το έγγραφο εργασία, έχω να πω πολλά πράγματα. Έχω σημειώσει δέκα σημεία, δεν έχω χρόνο όμως για να κάνω μια τέτοια παρουσίαση. Και γι' αυτό είμαι σε δύσκολη θέση και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα ε, να περιγράψω αυτά που έχω να πω. Τα έγγραφα εργασία και το πρώτο και το δεύτερο μέρο των έγγραφων εργασία είναι πολύ χρήσιμη παρουσίαση του ιστορικού και ε, των πολιτικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια. Το πρόβλημα με τα έγγραφα εργασίας είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώ την έγγραφη της Επιτροπής που για μας αποτελεί το σημείο σύγκρισης για αυτό το θέμα. Τα προβλήματα λοιπόν δεν αφορούν τα έγγραφα εργασίας αυτά καθεαυτά. Αλλά θεωρώ ότι λείπει ένα σχόλιο για την διεθνή στρατηγική ασφάλειας της Επιτροπής. Νομίζω ότι ε, είναι φυσιολογικές οι δυσκολίες που έχω, αλλά τι να σας πω, δεν έχω χρόνο τώρα για να τα περιγράψω τα σημεία που θεωρώ ότι λείπουν από τα έγγραφο εργασίας. Στις τροπολογίες μου θα προσπαθήσω να εξηγήσω τις ελλείψεις που διαβλέπω. Τι να σας πω, δεν έχω χρόνο να σας μιλήσω για θέματα ουσίας. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Το ξέρουμε. Αλλά πρέπει να είσαστε πολύ ε, περιεκτικοί. Κύριε Γιακολ, κύριε Γιακολίνο, και εσείς να είσαστε σύντομος. Θα ήθελα να πω ότι τα δύο έγγραφα εργασίας είναι πολύ καλό σημείο κίνησης. Όπως είπε και ε, ο κύριος Μπορσελίνο, η κυρία Μπορσελίνο, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μεταναστευτικές ροές, το έγγραφο αυτό θα λάβει τελική μορφή, διότι μην ξεχνάτε ότι εμείς ε, έχουμε να δεχτούμε ορδές μεταναστών στην Λαμπετούζα και τη Σικελία. Και τα δύο έγγραφα, και το έγγραφο Μπορσελίνο και το έγγραφο Αλφάνο, αφορούν θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο ε, συνεκτικοί και συνεπείς για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Κυρία Μπορσελίν, ας το αφήσουμε. Αν είναι για 30 δευτερόλεπτα δεν μπορώ να το κάνω. Ας το αφήσουμε. Εν πάση περιπτώσει η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα σύντομη. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε επιθεμάτων όπως εξετέθησαν και να πω για άλλη μια φορά ότι αυτό είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, το πρώτο βήμα. θα ήθελα να πω ότι και η έκθεση Σόνια Αλφάνο είναι εξίσου σημαντική. Πρόκειται για συμπληρωματικές εκθέσεις σε σχέση με θέματα που άπτονται της ασφαλείας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε, ε, να, αναβάλουμε τη συζήτηση έτσι ώστε να γίνει περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου. Η κυρία Μπορσαλίνο λέει κάτι εκτός... Ε, μικροφόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί έγινε μια πρώτη συζήτηση του εγγράφου εργασίας και με τη συνεργασία του Συμβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Θα το δούμε στην επόμενη συνεδρίαση. Τελευταίο σημείο σήμερα το πρωί, το υπαριθμό 12 συμμετοχή της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Η κυρία Ντέμπορα Σερακιάνη σε σχέση με τη συμμετοχή της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Ταξικομανίας είναι συντάκτρια θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία έχει οριστεί μέχρι αύριο στις 13 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και η σύσταση θα ψηφιστεί στις 2 Μαΐου. 2 Μαΐου. Ας ακούσουμε. Η κυρία Σεράκη. Grazie Presidente, cercherò di essere telegrafica. Come ricordava lei, si tratta del progetto... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Είναι ένα σχέδιο ψηφίσματο για μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία τη Κροατία για τη συμμετοχή τη Δημοκρατία τη Κροατία στην ε, λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την παρακολούθηση τη ε, τοξικομανία και των ναρκωτικών. Ένα κέντρο το οποίο βρίσκεται στην Λισαβόνα βασίζεται σε ένα κανονισμό του Φεβρουαρίου του 1993 και ε, το, κέντρο αυτό συλλέγει στοιχεία για τα ναρκωτικά και για την τοξικομανία. Ο στόχος είναι η διάδοση των πληροφοριών και η βοήθεια προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών. Από τον, Ιούλιο του 1996 το Συμβούλιο έδωσε την στην Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις που κατέληξαν το 1999. Ε, έγινε η αναθεώρηση της συμφωνίας ε, για να είναι συμβατή με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτεμβρίου του 2009. Γιατί είναι σημαντικό για την Κροατία να αποτελέσει τμήμα του παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά. Η Κροατία βρίσκεται σε ένα σημείο διέλευση και διαμετακόμισης ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγούς τις χώρες κατανάλωσης γίνονται κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ε, στην Κροατία και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός θανάτων που φύλλονται στα ναρκωτικά έχει αυξηθεί στην Κροατία. Ο ρυθμός ε, ε, των κατασχέσεων μειώθηκε τα τελευταία χρόνια εκτός από την ηρωίνη που παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για την ε, καταπολέμηση των ναρκωτικών και ε, υπάρχει ένας κατάλογος με τις πρόδρομες ουσίες ε, οι οποίες πρέπει να συνδυάζονται με το κοινοτικό κεκτημένο κατά το δεύτερο ήμιση του 2012 ή πρώτο ήμιση του 2013 πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πληροφορίες από την Κροατία για τα θέματα αυτά και επίσης είναι σημαντικό να μπορεί να επωφεληθεί η Κροατία από τη δουλειά που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και πρέπει να μάθουν για τις κοινέ πρακτικές υπάρχουν για την τοξικομανία και για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσα να είμαι περισσότερο σύντομη. Ευχαριστούμε κύριε Σερακιάνη. Ήσασταν πολύ σύντομη. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς ε, που έμειναν λίγο περισσότερο μαζί μας και έχουμε πολύ λίγο χρόνο για συζήτηση. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Όχι. Ο κύριος Σόκορ, σας παρακαλώ όλους να είστε πολύ σύντομοι. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα μιλήσω ουγγρικά. Θα ήθελα απλά να κάνω μία παρατήρηση. που αφορά ένα σημείο της έκθεσης. Η Κροατία αναφέρεται ως μια χώρα σε μετάβαση. Νομίζω ότι λέτε ότι υπάρχει λίγη κατανάλωση. Αν δείτε όμως τους αριθμούς είναι σαφές ότι η κατανάλωση στην Κροατία δεν είναι τόσο αμεληταία. Ίσως λοιπόν να μην λέμε ότι είναι μια ε, χώρα σε μετάβαση. Μια χώρα σε μετάβαση δείχνει χώρα που ανήκει σε άλλη κατηγορία. Γνωρίζω ότι ορισμένε χώρε ε, σε ένα ορισμένο πολιτικό πλαίσιο επιμένουν σε ορισμένε έννοιε. Οι χώρε σε μετάβαση είναι ορισμένε και νομίζω ότι πρέπει να βασιζόμαστε στα στοιχεία. Τι παρουσιάζουν τα στοιχεία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τάνακα, ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά στη θέση της Φρανσίσκα Κέλλερ ε, που είναι σιώδης συζητητής και μου ζήτησε να σας κάνω μια σύντομη παρέμβαση. Συμφωνούμε καταρχήν με τη συμφωνία, αλλά έχουμε μια παρατήρηση να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Και το άρθρο 5 της συμφωνίας τη γνώμη μα να έχει μια αλλαγή, θα κάνουμε μια τροπολογία, ώστε να προβλέπει την προστασία των δεδομένων. Κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτε άλλο, διότι η νομοθεσία στην Κροατία μοιάζει με εκείνη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συνεπώς, συμφωνούμε. Ευχαριστώ, κυρία Γκρίσβεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να είμαι τηλεγραφική και ελλειπτική, θα ήθελα να υπογραμμίσω απλά και μόνο ότι η ομάδα μας είναι απόλυτα ανοιχτή, αλλά και ενδιαφέρεται ε, από αυτό το νομοθετικό ψήφισμα που είναι συνέχεια διαπραγματεύσεων που θα καταλήξει σε συμφωνία που θα έχει δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα ένα σύστημα δικτύωσης και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της τοξικομανίας και της χρήσης των ναρκωτικών, δηλαδή τελικά καταπολέμηση όλων αυτών που μας απασχολούν, δηλαδή καταπολέμηση πάλι του οργανωμένου εγκλήματος και όλων των δεινών που πηγάζουν από αυτό και που χαρακτηρίζουν επίσης τη χρήση των ναρκωτικών. Τώρα, για τις αποχρώσεις χώρα μεταβατική, όχι με συγχωρείτε, χώρα διέλευσης ή χώρα σε διέλευση είναι κάτι το οποίο έχει ληφθεί υπόψη, ε, έχει δίκιο ο συνάδελφος, και το δεύτερο είναι η πρόοδος της ε, Κροατίας εν ώψη της εισδοχής ε, στον ε, ευρωπαϊκό χώρο. Θα δω τώρα με τους συναδέλφους αν θα κάνουμε τροπολογίες, αλλά πρέπει να βιαστούμε, εφόσον λίγη προθεσμία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ. Και η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς υποστηρίζουμε την έκθεση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορεί να συμμετάσχει και η Κροατία στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών για πολλούς λόγους είναι σημαντικό να δίδεται αυτή η δυνατότητα. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να συνεισφέρει στο να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα στην Ευρώπη για τα θέματα αυτά. Δεν θέλουμε να ε, υπάρχουν κρυφά στοιχεία, θέλουμε να υπάρχει μια απομυθοποίηση και δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνεται αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως με τη συλλογή δεδομένων μπορούμε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, θέλω να πω ότι ε, ε, θέλουμε ε, να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνούμε με την πρόταση των πρασίνων Υπάρχουν ε, κάποιε διατάξει ε, σχετικά με τα, δεδομένα, με προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν ε, να συλλέγονται. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Πρώτη φορά ασχολούμαι με αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί κανείς. Πάντως με αυτό το πρώτο σχέδιο είμαστε προς το ικανοποιημένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ και όλους ε, εκείνους που δεν έλαβαν το λόγο για να μας ε, βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας νωρίτερα. Υπενθυμίζω ότι είναι μια συμφωνία μεταξύ της Κροατίας και του Παρατηρητηρίου Ναρκωτικών. Δηλαδή, ε, μόνο διαδικαστικές μπορούν να είναι οι τροπολογίες οι διαδικαστικές επαναλαμβάνω τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι αύριο 13 Απριλίου 12 η ώρα. Για το συγκεκριμένο αυτό θέμα λοιπόν διαδικαστικές τροπολογίες μέχρι αύριο στις 12. Κυρία Στερακάνη, θέλετε να λάβετε το λόγο για να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα σχόλια για την προστασία των δεδομένων. Στο σχέδιο το οποίο υποβάλαμε ε, ε, καθίσατε σαφές ότι εφόσον αρχίσει η Κροατία να συνεργάζεται με το παρατηρητήριο θα ακολουθεί όλες τις διατάξεις ε, του κανονισμού και σε σχέση με την προστασία των δεδομένων θα ισχύσουν οι κανόνες που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω το σχόλιο αυτό να καθησυχάζει ορισμένε από τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και θα περιμένω τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος. Θα ξεκινήσουμε το απόγευμα στις 3.